Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ας ξεκινήσουμε. Στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης ο, κύριο, ο εισηγητής, ο κύριος Όλη Ρίστενσεν για τις ε, τροπολογίες ε, για την έκθεσή του για το ενωσιακό πλαίσιο εταιρική διακυβέρνηση δεν θα μπορέσει να έρθει αλλά θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Ζαρκάς από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Έχετε το λόγο. Efectivamente, lo primero es pedir eh, excusas en nombre de nuestro reporter, pero está en una reunión importante en, en un país africano. ¿no? Ο, ο εισηγητής είναι σε πολύ ε, σοβαρή συνεδρίαση και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου. μου. Λοιπόν, κατά την άποψη του εισηγητή, η στιγμή, η χρονική στιγμή της συζήτησης έχει ήδη πάρει το δρόμο της μπόρεσε να γίνει σημαντική πρόοδος στο Στρασβούργο και έχει δοθεί μια επιπλέον προσπάθεια για τις οδηγίες. 53 ε, τροπολογίες βρίσκονται στο συμβιβασμό που συνέταξε ο εισηγητής και οι 18 που παραμένουν βρίσκονται στις ε, αιτιολογικές σκέψεις, πράγμα που δεν δημιουργεί αξεπέραστες δυσκολίες. Όπως συνήθως όταν μιλάμε για, τις, για τους συμβιβασμούς ε, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για τις πληροφορίες ε, και μια σειρά από άλλα θέματα τις κοινωνικές επιπτώσεις, το κοινωνικό συμβόλαιο, την ε, πρόσβαση στη διακυβέρνηση και μια σειρά από άλλα θέματα. Όπως γνωρίζετε ότι ότι μεταξύ του αρχικού σχεδίου του συντάκτη και των συμβιβασμών υπάρχει διαφορά. Λαμβάνονται υπόψη σε αυτές τις περιπτώσεις σε μια σειρά από στοιχεία που διευκολύνουν τις σχέσεις εργαζομένων και εργοδοτών γιατί αυτοί οι κανόνες της ε, οικονομικής ε, διακυβέρνησης στις επιχειρήσεις δεν πρέπει να δεν ωφελούν μόνο τους εργαζόμενους αλλά και τους εργοδότες. Έτσι λοιπόν είναι επωφελής και προς τις δύο πλευρές. Παρατάρα υπάρχουν προβλήματα στις τροπολογίες είναι η G και η L εξακολουθούν να έχουν προβλήματα. Επ' αυτόν θα επανέλθω δεδομένου ότι τα υπόλοιπα περίπου έχουν διευθετηθεί ο υποχρεωτικός χαρακτήρας ή ο μη υποχρεωτικός χαρακτήρας των μέτρων για την εταιρική διακυβέρνηση είναι ένας ε, προβληματικός τομέας. Σύμφωνα με τον ε, συντάκτη έπρεπε να είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Είχε συντάξει μια ε, συμβαστική τροπολογία που έκανε τη διάκριση μεταξύ των μεγάλων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπήρχαν κάποια μέτρα που επέτρεπαν ευελιξία ε, για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως, αυτή είναι η χειρονομία που έκανε ο εισηγητής. Και εν κατακλείδη, κυρία Πρόεδρε, η συμβαστική τροπολογία L έκανε ο εισηγητής μια προσπάθεια να προσεγγίσει σημαντικά τις άλλες ομάδες. Κυρίως όσον αφορά την χρηματοοικονομική συμμετοχή αν διαβάσετε πολύ προσεκτικά την τροπολογία, συμβιβαστική τροπολογία του κ. Κρίστιανσεν, θα δείτε ότι η πρότασή του είναι λογική. Υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στις αμοιβέ και στο είδος αυτό της, και στο είδος της ε, επιδότησης του, του ε, επιπλέον ποσού που δίνεται στους ε, εργαζομένους, στους υπαλλήλους. Πρέπει να υπάρχει μια, βάση, μια βάση για την αμοιβή των εργαζομένων που ονομάζεται μισθός. Ο μισθός θα πρέπει να ρυθμίζεται από μια συλλογική ε, σύμβαση ή με ένα θεσμικό τρόπο. Όμως ο εισηγητής θέλει να βρει ένα άλλο σημείο ισορροπίας. Αυτό είναι άλλο σημείο που εκρεμεί. Ο κ. Κρίστανσεν μου λέει ότι μέχρι την Παρασκευή είναι διαθέσιμος για να ε, επεξεργαστεί ακόμα περισσότερο κάποιες διατάξεις. Όμως μου λέει ότι όλοι δεσμεύονται για την ουσία του θέματος που είναι υποφελής για όλους και νομίζω ότι αν καταβάλουμε μία ακόμα μικρή προσπάθεια θα βρεθεί μια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πάρει το λόγο, η κυρία Χάρκινς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ε, αντικαθιστώ τον Φίλιπ Ντεμπάκερ που ταξιδεύει για ένα συνέδριο θέλει καταρχήν να ευχαριστήσει τον εισηγητή για τις συμβιβαστικές τροπολογίες και για την παραγωγική συνεδρίαση που έχει γίνει. Εξακολουθεί όμως να θεωρεί ότι είναι απαραίτητες κάποιες προσαρμογές. Πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην εταιρική διακυβέρνηση και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Επιπλέον θεωρεί ότι δεν υπάρχει μία προσέγγιση που να καλύπτει τα πάντα. Φερρυπίν, σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν διαφορετικές εθνικές δομές εταιρικής διακυβέρνησης, πράγμα που δεν φαίνεται πάντοτε στην έκθεση. Δεν θα πρέπει να επισημαίνουμε συγκεκριμένα ε, εθνικά ε, παραδείγματα όπως η συναπόφαση, όπως τη συμβαστική δίτα. Ε, Επίσης υπάρχουν οι εισηγμένες και οι μη εισηγμένες οι χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εδώ αναφέρεται ε, στη συμβαστική λύση G. Επίσης πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προσπάθεια στην καλύτερη ε, λειτουργία και στην συμμόρφωση ε, με τις διάφορες συστάσεις όπως ισχύει στη διάφορα κράτη-μέλη και μόνο σε τελευταία περίπτωση και μόνο αν χρειάζεται η θα πρέπει να, λαμβάνονται υπόψη τα νομικά δεσμευτικά ε, μέτρα. Και θα έρθει σε επαφή με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για να δοθεί οριστική μορφή στις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κύριο Τόμας Μάν. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ο κύριος Κρίστενσεν είναι ένας από τους βουλευτές εκείνους ε, που είναι πρόθυμοι να δεχθούν συμβαστικές προτάσεις. Αυτό λοιπόν είναι ήδη μια πολύ καλή προϋπόθεση. Και θα ήθελα να επενθυμίσω ότι στην έκθεσή του περί και ασφάλειας μπορέσαμε να επιτύχουμε συμφωνία. Και το ΕΛΚ μας στήριξε. Όσον αφορά το θέμα CSR, ε, αυτό ε, δεν εμπίπτει πλέον στη δική μας την αρμοδιότητα, αλλά εμείς είμαστε μόνο οι συντάκτες ε, γνωμοδότησης. Και εδώ λοιπόν τίθεται και πάλι το ίδιο θέμα που παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι τίποτα το καινούριο. Είχαμε δύο εκθέσεις του τότε συναδέλφου Μπάσολ Μέθιους, ο οποίος είπε ότι αυτό θα πρέπει να παραμείνει προαιρετικό, αυτή είναι η σαφή θέση του ΕΛΚ, παραμένει η επιλογή προαιρετική. Τώρα υπάρχει άλλη άποψη. Λένε όχι προαιρετικό, ε, δεσμευτικό. Αλλά σε τελική ανάλυση κάποιοι ε, θα πρέπει να ασχοληθούν με την πραγματικότητα που επικρατεί στις επιχειρήσεις. Τι σημαίνει υποχρεωτικά, γιατί θα μπορούσαμε ίσως να πούμε οι μεγάλες να εξαναγκαστούν όχι οι μικρές, ούτε αυτό όμως γίνεται. Και αν δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες έχουν του εμπειρογνώμονες οι οποίες μπορούν να ενημερωθούν. Κάνουν μάλιστα και διαφήμιση με όλα αυτά. Και γιατί όχι. Αυτές ε, ίσως θα μπορούσαν να συμμετέχουν περισσότερο. Αλλά πώς θα γίνει αυτό με την δυνατότητα ε, να στηρίζουμε τις υπεύθυνε πράξεις ε, υπάρχει πρόοδο και αυτό το επιθυμούμε και εμεί. Θέλουμε να πείσουμε τι επιχειρήσει και αυτό δεν μπορεί να γίνει επιτακτικά τώρα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο. Δεν ξέρω πόσες φορές εσείς ε, έχετε επισκεφτεί επιχειρήσεις. Ε, γνωρίζω κάποιους που πηγαίνουν σε επιχειρήσεις τη Δευτέρα και την Παρασκευή και θέλουμε να ενημερωθούμε. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά αυτό το σύστημα της ε, ενημέρωσης, όπω ανάλυση θα καταλήξουμε σε ένα σύστημα που θα είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ίσως μπορούμε να πούμε <clears throat> ότι πρέπει να καλύπτονται κάποιες προδιαγραφές έτσι ώστε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς. Αλλά αν γίνει αυτό θα πρέπει να είναι προαιρετικό. Αναγκαστικά δεν γίνεται. Όταν θα επιστρέψει λοιπόν όλοι από το ταξίδι του, νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Αλεσάνδρο, το επισήμανε ε, πολύ καλέ οι συμβαστικές προτάσεις, μπορούμε να τις δεχθούμε, αλλά αυτή η ιδέα του να υπάρχει και πάλι ε, επιτακτική ανάγκη κανονισμού, εξαναγκασμός, αυτό έχει αποτύχει. Δεν μπορούμε να πούμε κάθε έξι μήνες θα υποβάλουμε το ίδιο θέμα το οποίο κατά την άποψη της Κομισιόν απέτυχε. Κάθε έξι μήνες το ίδιο θέμα στην ημερήσια διάταξη και το Κοινοβούλιο πρέπει μετά να αγωνίζεται. Δεν γίνεται αυτό Νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει επανειλημμένα. Αυτό ότι πρέπει να υπάρχουν εκθέσει που διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατόπιν τούτου, Αλεσάνδρο, θα πρέπει το θέμα αυτό να το εξετάσουμε από κοινού με τον Όλε. Ο συνάδελφο Χάτσκιν πολύ σωστά είπε, τα θέματα αυτά είναι κέρια. Ε, Βεβαίω μπορούμε να πούμε α περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην ψηφοφορία. Νομίζω όμω ότι μέχρι τώρα στην Επιτροπή Απασχόληση πάντα ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε το συμβασμό. Έτσι λοιπόν το πράσινο φω δεν έχει γίνει κίτρινο και ελπίζουμε όχι κόκκινο φω όπου θα καταλήξουμε στο ότι πρέπει να γίνει μάχη. Εντάξει, αν θέλετε μάχη γιατί όχι. Αλλά το προαιρετικό στοιχείο είναι ένα πολύτιμο αγαθό και δεν είναι κάτι το οποίο απλά είναι μια ε, τυχαία παρατήρηση. Γι' αυτό λοιπόν αν διατηρήσουμε την διακριτική ευχέρεια επιλογής, αυτό θα είναι πολύ καλύτερο να πούμε σε επιχειρήσει. παρακαλώ να συμμετέχετε περισσότερο αλλά όπως σα είπα προαιρετικά. Και γι' αυτό το λόγο ε, εμείς θέλουμε να στηρίξουμε αυτή την έκθεση. Θα ήθελα και εγώ να πάρω το λόγο επ' αυτού. Ο κύριος Τόμας Μαν μόλις ανέφερε το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε ε, στην προηγούμενη έκθεση του κυρίου Ματιός εκτιμώ αυτά που θυμάστε αλλά και εμείς ως Επιτροπή μαζί και κατά τη συζήτηση μιας γνωμοδότης ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των διατάξεων στον τομέα της ε, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Εντυπωσιάζομαι που ο κύριος Τόμας Μαν χαίρεται για το ότι υπάρχει πιθανότητα να είναι προαιρετικές ενώ όπως ξέρουμε είμαστε σε μια εποχή που επιβάλλονται αυτόματα κυρώσεις. Άρα είναι ε, κάπως πλάγια, η, πλάγιος ο τρόπος επίτευξης του αποτελέσματος. Σε πάση περιπτώσει, όσον αφορά τώρα τον προαιρετικό αυτό χαρακτήρα, όλη η στρατηγική της Λισαβόνας έγινε με προαιρετικές διατάξεις και είδαμε το αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε ε, πρέπει να αλλάξουμε. Ο κύριος Τόμας Μαν λέει ότι το έχουμε ήδη συζητήσει και δεν πρέπει να επανέλθουμε. Βεβαίως, γιατί καμιά φορά μιλάμε για τα υφιστάμενες ανισορροπίες στην, Ευρω... στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, πρέπει να επανέλθουμε. Ε, ίσως μερικά πράγματα πρέπει να τα ξανακάνουμε. Πολύ συχνά μιλήσαμε για τα ευρωομόλογα, δεν ήταν δυνατόν, τώρα ίσως θα γίνουν δυνατά. Θα Έτσι αλλάζει το πλαίσιο και ίσως θα πρέπει και εμείς να αλλάζουμε. Και βρισκόμαστε σε μια τέτοιου είδους φάση υπάρχει και το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης που έχει σχέση με αυτή την ε, ε, κρίση. Ο εισηγητής έχει αναφέρει ε, κάτι που, το οποίο με ευαισθητοποιεί. Πρέπει να διακρίνουμε στις επιχειρήσεις και να μην τις βάζουμε όλες το ίδιο τσουβάλι. Πρέπει να συμβιβαστούμε, να συνεργαστούμε από κοινού, να συντάξουμε μία, ένα συμβιβασμό που θα υπάρχει ευελιξία που μπορούμε να έχουμε ως ε, νομοθέτες να δούμε πότε θα εφαρμόζεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας. Μπορούμε ας πούμε να αφήσουμε τις μικρομεσαίες αλλά να υποχρεώσουμε ένα μεγάλο, μια μεγάλη ομάδα και ίσως ένα μεγάλο όμιλο, αλλά ε, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την προοδευτική εφαρμογή αυτών των διατάξεων είδα με ε, ενδιαφέρον τις αγορές, ε, την, την μετοχή της Société Générale. Στα, στους Γάλλους είναι πολύ γνωστή. Η Société Générale ε, είχε αποτελέσματα πολύ λιγότερο καλά από αυτά που είχαν προβλέψει και ταυτόχρονα ανακοίνωσε ότι δεν θα δώσει μπόνους. Αυτό δεν ήταν επιβεβλημένο από τον νόμο, αλλά θεωρήθηκε από τις αγορές ως θετική ένδειξη. Ως νομοθέτες δεν θα πρέπει να αισθανόμαστε ότι περιοριζόμαστε από τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Η καλή διακυβέρνηση είναι αφού έχουμε πειραματιστεί με το προαιρετικό χαρακτήρα ε, μπορεί να δείξει ότι πρέπει να γίνει υποχρεωτική, κάποιες διατάξεις να είναι υποχρεωτικές ώστε να πετύχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Ο κύριος Κρότσμαν έχει εγγραφεί στον κατάλογο και κατόπιν κλείνω τον κατάλογο των ε, αγορετών και κατόπιν ε, αυτός που αντικαθιστά τον νησί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, πραγματικά με εντυπωσιάζεται με τις ικανότητες ε, που επιδεικνύεται ε, ως πρόεδρος γιατί όταν υπάρχει κάποια παραβίαση αυτομάτως επεμβαίνεται και μάλιστα κατηγορηματικά. Σήμερα λοιπόν το πρωί το θέμα μας είναι πώς θα απαλλάξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το Small Business Act, ε, με τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλες που τάσσονται υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ένα τέτοιο, μια τέτοια έκθεση δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κόστος θα προκαλέσει. Γιατί υπάρχουν μεγάλε επιχειρήσει όπω η BASF, οι οποίε επιστοποιούνται από το Ινστιτούτο Περικολογικών Τήρη Κολογικών Προδιαγραφών και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε, όταν είναι μεγάλη επιχείρηση, είναι αναγκασμένη να πιστοποιηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, να συγκεντρώσει στοιχεία από παντού. Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητε ενέργειε. Ακούσαμε τι σημαίνουν όλα αυτά από πλευρά δημοσίευση ισολογισμών. Εντάξει, τα δεχόμαστε, αλλά με μια τέτοια έκθεση, αν περάσει, καλείται κανείς να δώσει επιπρόσθετες πληροφορίες και ε, πρέπει να προσφέρει και συγκεκριμένο περιεχόμενο αναπληροφορία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι τεράστιο κόστος. Ε, ε, αν θέλετε να το κάνετε σε ολόκληρη την Ευρώπη, μπορώ ήδη τώρα να σας πω τι θα συμβεί. Αυτή η εταιρεία την οποία αναφέρατε εσείς, αυτή η μεγάλη εταιρεία, ε, έχει τις πληροφορίες, αν θέλει βέβαια να τις ε, δημοσιοποιήσει προαιρετικά, αυτό μπορεί να γίνει, αλλά αν πιστεύετε επίσης ότι σε εθνικό επίπεδο μπορείτε να επιτύχετε μία ρύθμιση, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, οι Γάλλοι πιστεύουν ότι πράγματι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης, ας γίνει λοιπόν εκεί, αλλά στη τελική ανάλυση ας μην ξεχνάμε ότι εφόσον υπάρχει μια ρύθμιση ισχύει για το σύνολο της Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν στηρίζω τον συνάδελφο κύριο Μαν και αν αρχίσουμε στηρίξουμε στι επιχειρήσει επιχειρήσεις και εκεί να προβαίνουμε σε διαφοροποίηση γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τίθεται το όριο Πού θα βάλουμε, τι το θέμα, πού θα βάλουμε το όριο, τους 250 υπαλλήλους, γιατί δεν υπάρχουν ε, μικρομεσαίες που να είναι μεγαλύτερες. Κατόπιν τούτου καταλήγουμε στο ότι όλα αυτά είναι πάγιες δαπάνες, επιπρόσθετο κόστος το οποίο προκύπτει και θα πρέπει πάντα να κοιτάμε την απόδοση και όχι τον κύκλο εργασιών. Ε, λόγω της ε, χρηματοπιστωτικής κρίση ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται η πρόοδος δεν ενδιαφέρει, δεν με ακούει τώρα, αλλά επαναλαμβάνω λόγω της χρηματοψητικής κρίσης ελοχεύει κινδύνος να ε, πέσουμε σε ύφεση. Η οικονομία λοιπόν θα επιβραδυνθεί, δεν θα υπάρχει ανάπτυξη και εμεί τι κάνουμε, ανταυτού επιβάλλουμε νέο κόστο στι επιχειρήσει. Και υπάρχει και κάτι άλλο και θα κλείσω την παρέμβασή μου. Οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει είναι εκτεθειμένε ε, στον διεθνή ανταγωνισμό. Μέσα στην Ευρώπη θέλουμε και μπορούμε να επιτύχουμε ε, ίσου όρου ανταγωνισμού. Αλλά δεν γίνεται όμω αυτό να το επιβάλλουμε ε, σε παγκόσμιο επίπεδο και εδώ συμφωνώ μαζί σα ότι αν θέλετε να συγκεντρώσετε στοιχεία για την προστασία του περιβάλλοντο, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο σε μία χώρα. Γιατί για μία χώρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά σας λέω, πρέπει να έχετε το, το βλέμμα στραμμένο σε παγκόσμιο επίπεδο. Και ξέρετε να σας πω και κάτι άλλο συνάδελφε πρόεδρε, ούτε η Κομισιόν το θέλει αυτό που προτείνει η έκθεση. Δεν σας διέκοψα. και επιτρέψτε μου να σας ζητήσω να μην αμφισβητήσετε την ουδετερότητά μου κατά την άσκηση της Προεδρίας. Προεδρεύουσα, φροντίζω για την ισότιμη κατανομή του χρόνου ομιλίας και για την καλή οργάνωση των εργασιών μας. Αυτό δεν είναι ασύμβατο με το γεγονός ότι μπορώ και εγώ να μιλήσω ως αγορητής και με αυτήν μου την ιδιότητα εκ μέρους των σοσιαλιστών είπα ότι είπα. Αν εσείς θεωρείτε ότι μόνος πρόεδρος μπορώ να πανεβαίνω, διαφορούμε, λυπούμε επί της ουσίας. Συμμετέχω εδώ και ως πρόεδρος και ως ομιλητρία. Το επεισόδιο θεωρείται λήξαν, ήθελα όμως να προβώ σε αυτήν την διευκρίνηση όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκώ την Προεδρία. Στόχο μου είναι η απόλυτη ουδετερότητα. Για να κλείσουμε, ε, δίνω την Προεδρία στον Αντιπρόεδρό μας. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόιτσμαν για τα σχόλιά του. Τα μέλη της Επιτροπής μας πρέπει να συνειδητοποιήσουν το εξής. Εμεί εδώ νομοθετούμε και μάλιστα αν διαβάσετε και το κείμενο και τις τροπολογίες θα διαπιστώσετε ότι νομοθετούμε ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο με την έννοια ότι πρόκειται περί πράσινης βίβλου δεν πρόκειται για νομοθετικό κείμενο Ουσιαστικά, ακόμη, τουλάχιστον, δεν νομοθετούμε με την πρώτη έννοια του όρου. Θέλουμε να συστήσουμε αν οι εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν και κατά πόσον. Κύριε Κρότσμαν, εσείς πώς διακρίνετε μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Αν δούμε την τροπολογία την οποία έχουμε ονομάσει με το γράμμα G, διαβάστε το κείμενο. Θα βρείτε εκεί την απάντηση. Μην αντιτίθεστε σε κάτι το οποίο δεν υπάρχει ακόμη. Διαβάστε το κείμενο του εισηγητή. Ο στόχος είναι να διακρίνουμε μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων. Και η Κομισιόν προσπαθεί να καταθέσει και κάποια σχετικά κριτήρια. Προσπαθούμε, λοιπόν, μεταξύ άλλων να δούμε ε, τι ισχύει στον τομέα. Για παράδειγμα, κάποιοι θελοντικοί κώδικες συμπεριφοράς μεταξύ επιχειρήσεων. Είμαστε λοιπόν πρώτον πυλών ε, δημιουργίας ενός πλαισίου, το οποίο κάθε χώρα θα τον θεωρηλοποιήσει με τον δικό της τρόπο. Ο κ. Ε, Μαν και άλλοι συνάδελφοι είχαν την καλή διάθεση να πούν ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε. Εμείς δίνουμε μια γνωμοδότηση, δίνουμε τη δική μας άποψη ως Επιτροπή. Βρισκόμαστε όντως ε, σε ένα σταυροδρόμι στην Ευρώπη. Μεγάλες ε, επιχειρήσεις, μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υιοθετούν αυτοβούλως κώδικες συμπεριφοράς, τους οποίους όμως εν συνεχεία δεν τηρούν. Ο εθελούσιος λοιπόν χαρακτήρας αυτών των κωδίκων για τι συγκεκριμένε εταιρείε που αποτελούν ένα συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη ε, δεν ξέρω αν οδηγεί πουθενά. Ζητάμε πολλά όταν ζητούμε από αυτέ τι επιχειρήσει να λειτουργήσουν καλύτερα. Πώ άλλωστε το κάνουμε με τι χώρε μα, τα κρατημέλη. Αυτό κάνουν οι Γερμανοί. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Γερμανία. Υπάρχει ένα αποδοτικό μοντέλο, το κράτο λειτουργεί, οι επιχειρήσεις λειτουργούν, υπάρχει διαφάνεια. Συνεπώ. Δεν βλέπω να πρόκειται εδώ για σοσιαλιστική επανάσταση. Ούτε ζητούμε να σε μια δημοκρατική επανάσταση. Ζητούμε διαφάνεια, ζητούμε περισσότερη διαφάνεια για τις επιχειρήσεις. Κύριε Άρκιν, κύριε Κρότσμαν, κύριε Μαν, θα ήθελα να συμφωνήσουμε ότι το κείμενο είναι πολύ πιο ευέλικτο αυτό πρέπει να το αναγνωρίσετε. Και σα ζητώ να δείξετε κι εσείς την ίδια ευελιξία. Να αποφύγουμε τι ακραίε θέσει που δεν οδηγούν από την άλλη πλευρά πουθενά. Υπάρχει ένα κυρίαρχο μοντέλο στην Ευρώπη, θέλω να ισχύσει παντού. Ζητώ από του Γερμανού συναδέλφου να ρίξουν μια ματιά στο τι γίνεται στην Γερμανία και να συναγράφουν τα δικά του συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Η Τζούρι είναι η αρμόδια επιτροπή. Η έγκριση, η ψηφοφορία στην Ολυμένη θα γίνει τον Μάρτιο. Συνεχίζουμε με ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε τι κάρτε σα όλοι. Αν κάποιο δεν έχει την κάρτα του, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Για να σα συμπεριλάβουμε στην καταμέτρηση. Η πρώτη έκθεση. Η πρώτη έκθεση είναι η έκθεση της ε, Καρίμα Μαντέλη για την, ε, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Λοιπόν, συμβιβασμητική πρόταση C. Ποιος είναι κατά? Να, Αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά έλεγχος επί της 46 Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε αν έχετε πρόβλημα με το μηχάνημά σας. Πέρας ψηφοφορίας. 16 υπέρ, 18 κατά, καταπίπτει. 47 καταπίπτει, συμβασμός D υπέρ, κατά, αποχές, α, έλεγχος. Ανοίγουμε για το D. Πέρας ψηφοφορίας. 31 Α, όχι, δεν ήταν και το 31 υπέρ, 4 κατά. Πολύ περίεργο. Είδα κάποιους να πάνε να κάνουν προς τα κάτω τον αντίχειρα. Α, εν συμβαστική D εγκρίθηκε. Ή e τώρα, συμβαστική Ή. E, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και συνεχίζουμε με το συμβαστική G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. MV8 υπέρ, κατά, έλεγχος για το MV8. Πέρας. Η 20 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Έλεγχος επί του 58. Πέρας. καταπίπτει. 20 κατά, 16 υπέρ. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 60. Χωριστή ψηφοφορία. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Καταπίπτει. Τροπολογία 61 χωριστή ψηφοφορία. Υπέρ του πρώτου μέρους. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. 63 υπέρ. Κατά. Έλεγχος επί της 63. Ένα, αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18, 19. <laughs> Δεν εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, δεν εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 δεν εγκρίνεται. Καταπίπτει. 67 υπέρ κατά ε, έναρξη ψηφοφορίας για την 67. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 68 υπέρ, κατά. Θα πρέπει να κάνω έλεγχο. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV31 καταπίπτει ε, συμβιβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 έχει αποσυρθεί 72 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει Συμβιβαστική I υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και προχωρούμε στην άλλη σελίδα. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. 81. Είναι, α, έχει καταπέσει. Υπέρ, 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Θα κάνω έλεγχο για την 83 υπέρ. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 84. Προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση. Καταπίπτει. θα ψηφίσουμε ως προσθήκη χωρίς την προφορική τροπολογία. Μόνο για αυτό το σκέλος, το κομμάτι της 84, τα έχετε στον κατάλογο. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Σε αυτό το μέρος της 84. Έλεγχος. Πρόκειται για μια προφορική τροπολογία. Είμαστε κατά. Δεν πρέπει να ψηφιστεί η προφορική τροπολογία. Θέλουμε να ψηφίσουμε το κείμενο χωρίς την προφορική τροπολογία. Αυτό προσπάθησα ακριβώς και εγώ να διευκρινίσω, λέει η Πρόεδρος. Ε, όπως γράφει στον κατάλογο ψηφοφορίας, αφού εγκρίθηκε η 83 δεν ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία, ψηφίζουμε απλώς την προσθήκη των σημειώσεων ε, που λέει notes κλπ. Μπορούμε λοιπόν να επαναλάβουμε για την 84, έλεγχος για την 84. Αρχίζει ψηφοφορία για την 84. Πέρας ψηφοφορίας. 27 υπέρ, 7 κατά, εγκρίνεται. «85 καταπίπτει, 86 είναι συμβατή, υπέρ της 86, κατά έλεγχος, έναρξη ψηφοφορίας για την 86». Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας, 25 υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. 87. Ψηφίζουμε. Δεν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εμπερδεύτηκα, λέει πρόεδρος. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 88 έναρξη. Οι συντονιστέ σας μου κάνουν σήμα. Πέρας. 16 υπέρ, 19 κατά, καταπίπτει. 89 υπέρ, κατά, καταπίπτει. 90 υπέρ, κατά. Αποχές, έλεγχος για την 90, έναρξη. Πέρας, 20 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 91 έλεγχος πέρας ελέγχου 15 υπέρ 21 κατά δεν εγκρίνεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά ε, αποχές κατά αποχές. Συμβιβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV18 καταπίπτει συμβιβασμός K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά θα ελέγξω την 97 έναρξη πέρας 20 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται 98 υπέρ κατά Καταπίπτει. 99. Αποσύρεται. 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. NV2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102. Καταπίπτει. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Συμβιβαστική θα ελέγξουμε, θα ελέγξουμε. 101 ε, έλεγχος. Πέρας. Είμαι σίγουρο ότι ε, δεν εγκρίθηκε με σημαντική διαφορά. Λοιπόν, δεν εγκρίνεται. Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και προχωράμε στο συμβιβαστική αίμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. Συμβιβαστική εν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά. Έλεγχος στην 116, νομίζω ότι δεν εγκρίθηκε, αλλά να δούμε. 116 ε, έναρξη. Πέρας. 19 υπέρ, 15 κατά, εγκρίθηκε. 117 υπέρ, κατά Αποχές εγκρίνεται. NV32 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική O. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV22 καταπίπτει. NV27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. Συμβασμός π. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται φτάνουμε στο 132. Καταπίπτει 133 υπέρ, κατά, θα κάνω έλεγχο για το 133. Έναρξη. Πέρας. 21 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. 134 υπέρ, κατά. Αποχές το ίδιο νομίζω, αλλά έλεγχο. 134 έναρξη. Πέρας. 20 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 137 χωριστή ψηφοφορία, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, Έλεγχος του δεύτερου μέρους της 137, έναρξη. Πέρας. 13 υπέρ, 23 κατά, δεν εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά. Αποχές, καταπίπτει. Συμβιβαστική Q, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 131 είναι συμβατή με την 138. Εγκρίθηκε 138. Η 139, αυτήν συζητώ λέει η πρόεδρος. Όχι. 139 όντως καταπίπτει. 140 144 αποσύρθηκε, 145 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 147 καταπίπτει, 148 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 150 έναρξη. Πέρας. 17 υπέρ, 20 κατά, καταπίπτει. 151 υπέρ, κατά. Αποχές, έλεγχος για την 151 έναρξη. Πέρας. 21 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Έλεγχος στην 155 έναρξη. Πέρας. 20 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV6 καταπίπτει. NV30 υπέρ, κατά, Αποχές, α, έλεγχος, έλεγχος, έναρξη. Πέρας. Δεκατρία υπέρ, 22 κατά, δεν εγκρίνεται. Σύμβιβας R υπέρ, ε, ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά, αποχές, Έλεγχος 160. Έναρξη. Κάποιος δεν ψήφισε. Πέρας ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 17 κατά. Εγκρίνεται. 162 είναι συμβατή με την 160 και 161 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι δεν εγκρίνεται, αλλά έναρξη ψηφοφορίας για την 162. Πέρας. 16 υπέρ, 21 κατά, δεν εγκρίνεται. Συμβιβαστική S. η 163 θα ψηφιστεί μετά. 164 υπέρ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική Z υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος έναρξη για την 168 πέρας 20 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται 169 υπέρ κατά έναρξη ελέγχου 169 έλεγχος Ένας ακόμα να ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 22 κατά, καταπίπτει. Ε, 170 υπέρ, κατά, αποχές, δεν εγκρίνεται. NV7, NV7 υπέρ, κατά, αποχές, δεν εγκρίνεται. NV10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 171-72 αποσύρθηκαν, 173. Να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. Συμβιβαστική τι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 176 υπέρ, κατά. Πρέπει να κάνω έλεγχο έναρξη. Πέρας. 15 υπέρ, 22 κατά, δεν εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, ε, καταπίπτει. 180 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. NV3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 182 καταπίπτει 190 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Έλεγχο στην 193. Έναρξη. Πέρας. 15 υπέρ, 22 κατά, καταπίπτει. 194 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. 194. Έλεγχος. Ένας ακόμα πρέπει να ψηφίσει. Κάποιος δεν έχει ψηφίσει. Πέρασε. Υπέρ. Α, όχι. 20 <laughs> υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. 195 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. NV18 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 198 καταπίπτει, 199 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. S, συμβαστική S, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οπότε τώρα αντικαθιστά το, την 163 από ό,τι μου λένε, οπότε προχωρούμε στο 203 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. 205 υπέρ. Κατά. Καταπίπτει. 206 υπέρ. Κατά αποχές καταπληκτή. Συμβιβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 210 υπέρ κατά αποχές ε, ε καταπίπτει. 211 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.16 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. NV16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.17 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. 2.18 αποσύρθηκε. 2.19 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος τη 219 έναρξη. Νομίζω ότι δεν εγκρίνεται, αλλά για να δούμε. Πέρας. 16 υπέρ, 21 κατά, δεν εγκρίνεται. 2,20 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2,21 υπέρ, κατά, αποχές καταπίπτει. 222. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 232 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 233 υπέρ κατά αποχές Καταπίπτει. NV23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.34 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για τη 2.34 έναρξη. Πέρας. 16 υπέρ, 21 κατά, δεν εγκρίνεται. 2.35 υπέρ. Κατά αποχές καταπίπτει 2.36 υπέρ κατά έλεγχος για τη 2.36 έναρξη πέρας 22 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται 2.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.39 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. 2.40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.41 υπέρ. Κατά. Αποχές καταπίπτει. 2.42 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, δεν εγκρίνεται. NV14 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 από την Επιτροπή ΦΑΜ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ Κατά. Αποχέ ε, κατά αποχές καταπίπτει. 6 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται 12 δεν εγκρι... Ε, καταπίπτει 13 υπέρ κατά αποχές δεν εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική A υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά. Έλεγχος για την 21, έναρξη.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, θα, έλεγχος για την 31, έναρξη. Πέρας ελέγχου. 22 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται. 32 είναι συμβατή, υπέρ λοιπόν. Κατά, και πάλι δεν διακρίνω έλεγχος για την 32 πέρας νομίζω ότι εγκρίθηκε αλλά για να δούμε όχι δεν εγκρίθηκε 16 υπέρ 21 κατά 33 συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 καταπίπτει 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 37 από τη ΦΑΜ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 ΦΑΜ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και, και τέλος θα ψηφίσουμε την τελική έκθεση έναρξη. Δύο δεν ψήφισαν. Ένας ακόμα πρέπει να ψηφίσει. Πέρας ψηφοφορίας. 36 υπέρ, 2 κατά, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για τη σκληρή δουλειά που έκανε. Oh, the next vote is, um, Τώρα θα ψηφίσουμε λοιπόν για την επόμενη έκθεση του κυρίου Γκίγκολτ, ε, καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συντηρισμού σε αφορά το ρόλο των εργαζομένων. Ε, καταρχήν για την ε, τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 26 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 27 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 28 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 29 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές ε, καταπίπτει 32 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει η ε, συμβαστική α υπέρ κατά αποχές καταπίπτει μισό λεπτό όχι όχι εγκρίνεται λάθος τρελάθηκα λοιπόν πάμε στην συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Για την D πάμε συμβαστική E υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Ε, η νομική 2, jury 2 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, jury 3 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, η 44 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, η 45 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, 46 υπέρ κατά, αποχές καταπίπτει, 47 καταπίπτει, 48 καταπίπτει, 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 50 καταπίπτει, η συμβαστική G υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η ε, Τζούρι Νομική Επιτροπή 5 υπέρ κατά αποχές Συγγνώμη, επανέρχομαι στην Τζούρι 5, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική L, υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΦΑΜ 4 καταπίπτει μέχρι την ΦΑΜ 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική H υπέρ, κατά, Μισό λεπτό. Ε, συγγνώμη, τώρα όταν μετακινήσετε και ψηφίζετε κιόλα, ε, με, δυσκο... με δυσκολεύει πάρα πολύ. Μήπω μπορείτε, σα παρακαλώ, τουλάχιστον να κάθετε για να βλέπω κι εγώ πώ ψηφίζετε. Έχετε καλοσύνη, παρακαλώ, να καθίσετε. Δεν βλέπω αυτού που σηκώνουν τα χέρια τους, λυπάμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, συμβιβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 64 υπέρ κατά αποχές, μισό λεπτό, ε, θα το επανελέγξω. Η 64, δεν το είδα καλά, ε, άρχεται η ψηφορία για την 64. Έκλεισε. 23 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. Η επόμενη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 66 καταπίπτει, η 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 68 υπέρ, κατά, αποχές, καταπίπτει. Πάμε στην 69. Εδώ υπάρχει προφορική τροπολογία. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ε, Έλεγξα την 71. Για το 71 ψηφίζουμε. Ε, καταπίπτει ε, χωρίς καμία αμφιβολία έκλεισε η ψηφοφορία νομίζω είναι σαφές το αποτέλεσμα Δύο υπέρ 40 κατά κάτι δεν πήγε καλά εδώ συμβιβαστική α υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται η 74 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 80 υπέρ κατά αποχές, ε, συγγνώμη, αλλά σας παρακαλώ να κάθεστε αν έχετε καλοσύνη. Δεν μπορώ να βλέπω πώς ψηφίζουν οι υπόλοιποι. Το 80 παρακαλώ υπέρ, κατά. Ε, πρέπει έτσι κι αλλιώς να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 80 παρακαλώ. Σα ε, Σας παρακαλώ ε, να μην κάθετε κανείς όρθιος στη μέση ε, μέχρι να τελειώσει ψηφορία γιατί σας λέω δεν βλέπω πώς ψηφίζουν οι υπόλοιποι και γίνεται πρόβλημα. Λοιπόν, Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο. Η συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 86 υπέρ κατά εγκρίνεται η τροπολογία ΦΑΜ 1 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται η ΦΑΜ 2 υπέρ η ΦΑΜ 2 ξαναψηφίζουμε για την ΦΑΜ 2 Παρακαλώ ποιοι είναι υπέρ της ΦΑΜ 2 κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Η 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Η 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Ε, όχι, όχι, αυτή εγκρίθηκε. Η 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει. Η 5. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 7 ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές καταπίπτει. Η 8 υπέρ, κατά, αποχές καταπίπτει. Η 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ, κατά, αποχές καταπίπτει. Η 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η 12 καταπίπτει και πάμε τώρα στην 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 17 υπέρ κατά ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 17 παρακαλώ Λοιπόν, ε, η ψηφορία ξεκινάει για την 17 Έκλεισε η ψηφοφορία. Καταπίπτει λοιπόν. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 19 υπέρ, κατά αποχές καταπίπτει. Η 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές ε, καταπίπτει. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 23, το 24 μπερδεύτηκε η πρόεδρος, υπέρ κατά, αποχές ε, εγκρίθηκε. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφορία για το τελικό αποτέλεσμα. Ψηφίζουμε παρακαλώ. The vote is closed. 41 in υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια ε, στον εισηγητή. και τώρα σχέδιο γνωμοδοτησής Κοφεράτη. Ψηφίζουμε. Πρόταση οδηγίε Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τι προποθέσει εισόδου και διαμονή υπηκών τρίτων χωρών για εποχική απασχόληση. it's an exception yeah. to our rule that yeah. deletions come first. Okay. Right. Um, 86. 86 αποσύρθηκε συμβαστική J αντικαθιστά τη 14 ε, και 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 καταπίπτει παίρνουμε στη συμβαστική και, και υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. L συμβαστική. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Με συγχωρείτε. Η L υπέρ. Ξανά. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 και 94 δεν έχουν γίνει αποδεκτές. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 102 υπέρ κατά αποχές καταπίπτει 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 105 δεν είναι αποδεκτή. Συμβαστική N υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 106 μη αποδεκτή. Ο όμικρον υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 109 ε, μη αποδεκτή. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...153 έχει αποσυρθεί... 162 είναι προφορική για να αντικαταστήσει τις λέξεις, ε, μερικές λέξεις υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος, έναρξη ψηφοφορίας για την 162. Ψηφίζουμε λοιπόν είπα πέρας ψηφοφορίας. ...23 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται. Συμβαστική T, ταφ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική U υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άρθρο 17. Ο εισηγητής προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική πι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. D. Συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35 υπέρ. Έλεγχος για την 34. Νομίζω ότι, ήταν, ότι εγκρίθηκε, αλλά ψηφίζουμε. την 34. Πέρας. 25 υπέρ, 18 κατά εγκρίνεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ίδιο. 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 έως 42 να τις δούμε μαζί αυτές 37 έως 42 όχι α είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική βή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά 44 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Βλέπω χέρια πάνω κάτω. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 44 πέρα ψηφοφορία, 25 υπέρ 18 κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Συμβαστική β, β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε διάφορες που έχουν αποσυρθεί. 50-52 μη αποδεκτή. 3. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53 υπέρ. Συμβατή. Κατά. Αποχές. καταπίπτη. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Α, όχι, με συγχωρείτε, καταπίπτει. 55 καταπίπτει το ίδιο, 56 το ίδιο και 57. Πάμε στη συμβαστική C. Υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός για την σε, συμβαστική σι. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφορίας. Να σίγουρος ότι έχει εγκριθεί, αλλά να δούμε πέρας ψηφορίας. Α, 41 υπέρ 2 κατά. Ναι, μια μικρή πλειοψηφία. 61 μη αποδεκτή. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική F υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές. Καταπίπτει 7 υπέρ. Α, ε, ηλεκτρονική ψηφορία για την 6. Είδατε, μόλις με το που δίστασα στη φωνή μου, την 6 ψηφίζουμε. Πέρας. 24 υπέρ, 19 κατά, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 αποσύρεται. 71 υπέρ, κατά, εγκρίνεται που θέλει να διάρθει τις προηγούμενες. Υπέρ. Κατά. Υπέρ. Ξαναψηφίζουμε για την 74. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καταπίπτει λοιπόν συμβαστική G. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική... Α, η 10. Έχουμε τη 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ενδέκατη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I Ι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά έλεγχος για την 84. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 22 υπέρ, 21 κατά. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Να το δούμε ηλεκτρονικά. Για την 85 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφορία 21 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. Το αντίθετο. Καλά κάναμε και ελέγξαμε και ψηφίζουμε επί του συνόλου έναρξη ψηφορίας. The vote is closed. πέρας ψηφορίας. 39 υπέρ, 3 κατά μία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Κοφεράτη. Κλείνουμε λοιπόν με τις ψηφορίες και περνούμε διασωκέ για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση εργαζομένων στον κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από φυσικούς παράγοντες και συγκεκριμένα σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες. Διακόπτουμε για λίγα λεπτά για να φύγουν κάποιοι, να έρθουν κάποιοι άλλοι και να δώσουμε και τη θέση της στην εισηγήτρια. Όσοι να φύγουν παρακαλώ να αποχωρήσετε το συντομότερο δυνατόν. Ξεκινάμε λοιπόν για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παρακαλώ, καθίστε. Η οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. η οδηγία για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Παρακαλώ καθίστε για να μπορώ να δώσω το λόγο στην κυρία ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα Πρόεδρος, δυστυχώς δεν μπορούμε να ακούσουμε την εισηγήτρια την κυρία Μωράν Σαρτιέ Παρακαλώ, αν θέλετε να συζητήσετε, να βγείτε. Λοιπόν, κυρία Μωράν Σαρτιέ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Μια πολύ λεπτή κατάσταση. Το σημαντικό θέμα αφορά την υγεία των εργαζομένων, η οποία, οι οποίοι υπόκεινται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με το θέμα της υγείας των εργαζομένων και αυτό ε, εξαιρεί οτιδήποτε μπορεί να έχει συμπεριληφθεί σε αυτή την οδηγία και η οποία δεν αφορά κατά τη στενή έννοια την υγεία των εργαζομένων. Οποιαδήποτε παρατήρηση που δεν αφορά την υγεία των εργαζομένων οι οποίοι υπόκεινται σε πεδία ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι εκτός της το πεδίο της οδηγίας. Δεύτερον, έλεγα ότι η κατάσταση είναι λεπτή, το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα κυρία Πρόεδρε, επειδή το 2004 υπήρξε μια οδηγία για την υγεία των εργαζομένων που υπόκεινται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, η οποία αποδείχθηκε μη εφαρμόσιμη αν δεν θέλαμε να αποκλειστεί η χρήση της ηλεκτρομαγνητικής, της ηλεκτρομαγνητικής απεικόνησης, η οποία είναι απαραίτητη. και η ισχύς παρατάθηκε μέχρι τις 30 Απριλίου 2012. Επιτέλους βρισκόμαστε στο τέλος της ε, περίοδου της παράτασης της οδηγίας του 2004 και μπορώ να ανακεφαλαιώσω την κατάσταση ως εξής. Είμαστε υποχρεωμένοι να εγκριθεί ένα κείμενο πριν από τις 30 Απριλίου του 2012 αν δεν θέλουμε να ξαναβρεθούμε στην ίδια δυσκολία και να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ε, ιατρική χρήση της ε, ε, ηλεκτρομαγνητικής απεικόνησης. Η κατάσταση σήμερα έχει ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε διαμακρών, διαβουλεύθηκε με όλους τους εταίρους. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η εργασία που έγινε σε βάθος χρειάστηκε χρόνο και γι' αυτό ακριβώς το σχέδιο οδηγίας που από καιρό αναμενόταν στην Επιτροπή έφτασε με καθυστέρηση, με κάποια καθυστέρηση. Εκ παραλίλου γνωρίζω ότι σε επίπεδο του Συμβουλίου οι εργασίες που αυτή τη στιγμή γίνονται υπό την Πολωνική Προεδρία ενημερωτικά και βεβαίως έχουμε συντονιστεί με το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες διότι θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στο Συμβούλιο υπάρχει σήμερα μία μειοψηφία κρατών μελών που έχουν αντιρρήσεις για την ε, εξαίρεση της, ε, ε, της μαγνητικού συντονισμού. Είναι η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Λιθουανία, η Γερμανία και η Τσεχία. Σήμερα λοιπόν μας έχουμε, πρέπει να βρούμε ένα κείμενο που θα ισορροπεί αφενός με την υγεία αυτών οι οποίοι εργάζονται σε αυτά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που μας απασχολεί όλους, αλλά από την άλλη πλευρά την απαραίτητη χρήση της απεικόνησης μαγνητικού συντονισμού που χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αύριο μπορεί να είμαστε εμείς ο ασθενής, το παιδί μας, ε, ο σύντροφός μας, ε, ένας συγγενής μας. Και δεν θα πρέπει να φανταστούμε ότι υπάρχουν άλλες τεχνικές πέρα της μαγνητικής τομογραφίας που θα αντικαταστήσουν κάποιες ε, ιατρικές εξετάσεις. Σήμερα αυτές οι τομογραφίες είναι απολύτως απαραίτητες για την παρακολούθηση της εξέλιξης κάποιων ασθενών, για, την νευρο για τις νευροεπιστήμες, για τα εγκεφαλικά ε, επεισόδια, για την παρακολούθηση της εξέλιξης καρκίνων, για την παρακολούθηση της εξέλιξης ασθενειών όπως το Αλτσχάιμερ, ή εν πάση περιπτώσει οι, οι ασθένειες που οφείλονται στην γύρανση του πληθυσμού ε, βρισκόμαστε λοιπόν στο επίκεντρο όχι μόνο του θέματος της υγείας των εργαζομένων αλλά και στο επίκεντρο του θέματος της δημόσιας υγείας ε, και της υγείας μας. Η δουλειά της Επιτροπής λοιπόν λαμβάνει υπόψη της την απαραίτητη αυτή προσαρμογή της οδηγίας του 2004 ώστε επιτέλους να μπορέσουμε να εποφεληθούμε εξίσου και από την προστασία των εργαζομένων αλλά και να ε, χρησιμοποιούμε τις μαγνητικές απεικονίσεις. Υπάρχει μια δεύτερη εξαίρεση, μια δεύτερη παρέκκληση που ε, περιλαμβάνεται στο σχέδιο αυτό οδηγίας που αφορά την άμυνα και σε αυτή, αυτή την περίπτωση σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα. Αυτή η νέα οδηγία, αυτό το νέο σχέδιο κειμένου μας έδωσε τη δυνατότητα να ε, εργαστούμε εξαιρετικά συντονισμένα με τους σκιώδεις εισηγητές της Επιτροπής Απασχόλησης, δεδομένου ότι οργανώσαμε μια σειρά από συνεδριάσεις με βάση την αρχή ότι εμείς μεταξύ μας επιθυμούσαμε να γίνει γνωστό να μοιραστούμε τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες και από την Επιτροπή και το Συμβούλιο συγκεντρώθηκαν επιστημονικές πληροφορίες έτσι ώστε όλοι οι σκιώδεις εισηγητές να μπορούν να δουλέψουν πολιτικά και στις πολιτικές τους ομάδες και να έχουν τις ίδιες βασικές πληροφορίες. Θέλω να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές οι οποίοι ασχολήθηκαν με την οδηγία αυτή έδειξαν ένα ε, πνεύμα συνεργασίας, ε, επιμέλειας, ε, συντονισμού και κυρίως ασχολήθηκαν σοβαρά. Ο συντονισμός που έχει ήδη ξεκινήσει και πρέπει να πω ότι με τον ε, συνάδελφο και φίλο τον Αλεσάνδρο Σέρκας ήδη κάναμε προγραμματισμένη δουλειά με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα για το θέμα αυτό. Ήδη είχαμε και επαφές με αυτούς οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της υγείας ε, ε, σε περιβάλλον μαγνητικού συντονισμού με ασθενείς, με γιατρούς, με κατασκευαστές. Κάναμε μια ευρεία διαβούλευση η οποία αυτή τη φορά θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε μια οδηγία η οποία θα είναι λειτουργική, θα είναι άξια του ονοματός της και η οποία θα κάνει ε, περήφανη την Ευρώπη, γιατί εγώ δεν αισθάνομαι καμία υπερηφάνεια που πρέπει να ξαναδουλέψουμε μια οδηγία του 2004, η οποία δεν είναι εφαρμόσιμη, χωρίς να εγκαταλείψουμε ένα μεγάλο επίτευγμα της υγείας. Στις αρχές εβδομάδες, ε, στη, στην αρχή της εβδομάδας παραβρέθηκα στη συνεδριά της Επιτροπής Περιβάλλοντος για να παρακολουθήσω τη συζήτηση από αυτής της οδηγίας. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος επιδεικνύει το ίδιο πνεύμα με μας. Ε, άκουσα μια έντονη έκκληση από έναν ε, συνάδελφο στην Επιτροπή να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους συναδέρφους των χωρών οι οποίοι διαιρωτώνται για την εξαίρεση κάποιων τομέων. τομέων. Είναι ευθύνη όλων μας, θεωρώ, να προχωρήσει αυτή η οδηγία. Πρέπει να σας πω ένα πράγμα, ότι σήμερα αν στη μαγνητική απεικόνηση δεν γνωρίζουμε, αν δεν γνωρίζαμε αν, πώς να προωθήσουμε την οδηγία του 2004, μην φανταστείτε ότι το σκάνερ μπορεί να υποκαταστήσει τη μαγνητική ε, απεικόνηση. Είναι πολύ έχει πολύ περισσότερη εκτινοβολία, άρα τίθενται πολύ μεγαλύτερα ερωτήματα για την επίπτωση στην υγεία και των ασθενών και των εργαζομένων, αλλά αφετέρου η μαγνητική απεικόνηση είναι απολύτως αναντικατάσταση, είναι μια εξέταση απολύτως αναντικατάσταση για τις παθήσεις που ανέφερα προηγουμένων τις άνοιες, τη σκλήρηση κατά πλάκα, τις νευρολογικές παθήσεις και μια σειρά από άλλες. Βεβαίως θέλω να σας πω ότι η δουλειά η οποία κάνουμε σε αυτό το πνεύμα κινείται και υπολογίζω ότι όλοι οι εισηγητές θα μπορέσουν να βοηθήσουν να πετύχουμε αυτό το διπλό αποτέλεσμα. Όφελος προς τους ασθενείς αλλά και διατήρηση της ε, υγείας των εργαζομένων οι οποίοι υπόκεινται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε εδώ για να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων. Ε, ευχαριστώ η κυρία Χάπτη και μετά κυρία Λίν. Η κυρία Ράπτη και μετά η κυρία Λίν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, η κυρία Σαρτιέτα είπε τόσο ωραία που θα μπορούσα να πω μα συμφωνώ και πάμε παρακάτω. Ε, την ευχαριστώ για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει μέχρι τώρα. Μας έχει δώσει ένα εξαιρετικό κείμενο βάσης για να εργαστούμε και επίσης πρέπει να σημειώσω τη διαφάνεια με την οποία εργάστηκε. Όλα τα δεδομένα, όλες τις πληροφορίες που είχε και φρόντισε να βρει, α, τις μοιράστηκε αμέσως με τους σκιώδεις. Αυτό διευκολύνει εξαιρετικά τη δουλειά μας, σε σημείο που να, θέλω να είμαι αισιόδοξη ότι αυτή η νέα προσπάθεια που κάνουμε θα έχει επιτυχία. Και για να έχει επιτυχία το ξέρουμε όλοι ότι το στοιχείο της επιτυχίας είναι ένα. Να μπορεί η οδηγία να εφαρμοστεί. Ε, υπάρχουν βεβαίως κάποιοι προβληματισμοί. Τους ανέφερε και η εισηγήτριά μας. Είναι προβληματισμοί τους οποίους μοιραζόμαστε. Ε, είναι προβληματισμοί που πρέπει να συζητήσουμε για να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το κείμενο ώστε να μπορεί ε, όπως είπα προηγουμένως οι διατάξεις του να εφαρμοστούν προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Ε, ξέρω πολύ καλά όπως όλοι μας ότι για πολλές εφαρμογές η τεχνολογία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι αναντικατάστατη. Η περιγραφή που έκανε η Ελιζαμπέτ τα λέει όλα. Τώρα, η οδηγία αναφέρεται στις άμεσες επιπτώσεις από την έκθεση των εργαζομένων στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ξέρω πως εδώ υπάρχουν οι μακροχρόνιες και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις ε, γνωρίζω επίσης ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία επιστημονικά τεκμηριωμένα που να αποδεικνύουν μακροχρόνιες επιπτώσεις από την έκθεση των εργαζομένων στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Αλλά, από την άλλη πλευρά, η ιατρική έρευνα συνεχώς προχωρά, βελτιώνεται και η τεχνολογία των συσκευών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και αυτή με τη σειρά της εξελίσσεται. Με βάση αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις ώστε ε, να κάνουμε τις αλλαγές στην ομοθεσία που ενδεχομένως να χρειαστούν. Στο ίδιο πνεύμα θα ήθελα να αφαιρθώ και στη διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στις επιπτώσεις στην υγεία και στις επιπτώσεις στην ασφάλεια. Ε, δεν νιώθω πάρα πολύ άνετα με αυτή τη διάκριση. Ε, νομίζω ότι για το θέμα θα πρέπει να υπάρξει μια αναφορά. Προβλέπουμε βεβαίως τις αναγκαίες προφυλάξεις. Απ' την άλλη πλευρά χρειαζόμαστε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι άμεσες επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δεν θα μετατραπούν σε μακροχρόνιες. Ε, πηγαίνω έτσι στη λεπτομέρεια γιατί όλοι μας έχουμε στο μυαλό μας τους ασθενείς που πρέπει να γίνουν καλά και που είναι πολύ χρήσιμα τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία αλλά πρέπει να έχουμε και στο μυαλό μας τους εργαζομένους και τους κανόνες προστασίας στην πρόταση οδηγίας προβλέπονται και κάποιες εξαιρέσεις για κατηγορίες εργαζομένων. Καταλαβαίνω εδώ ότι τόσο τα επιχειρήματα υπέρ, καταλαβαίνω και τα υπέρ και τα κατά. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε στα κράτη τη δυνατότητα να εφαρμόσουν κάποιες αυστηρά περιορισμένες εξαιρέσεις έχοντας όμως πάντα υπόψη μας, σε αυτό επιμένω συνεχώς, την επιστημονική τεκμηρίωση και αιτιολόγηση ε, για τους αυστηρότερους κανόνες για τους εργαζομένους σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν θα ήθελα, για παράδειγμα, ε, να, μία μη τεκμηριωμένη προσέγγιση να αιτιολογεί α, λιγότερες ώρες εργασίας, για παράδειγμα και αυτό το λέω γιατί νομίζω ότι οι εργαζόμενοι ε, δεν πρέπει, να προστατεύονται, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να βρίσκουν καταφύγιο εντός εισαγωγικών σε ε, δικαιολογίες εύκολες και μη τεκμηριωμένες. Θέλω επίσης να τονίσω, έχοντας στο μυαλό μου αυτούς που ενδεχομένως αμφισβητούν την επιλογή των οριακών τιμών έκθεσης, τις οποίες χρησιμοποιούμε στην δουλειά μας, πως είμαστε υποχρεωμένοι, ε, έτσι τουλάχιστον το αισθάνομαι εγώ, να δεχτούμε έναν, τα δεδομένα που μας δίνει ένας διεθνός και ευραίος γνωστός επιστημονικός φορέας. Ε, τον λέω στα αγγλικά, International Commission on ionizing Radiation Protection. Είναι ε, η Διεθνής Επιτροπή, αν το λέω σωστά, των μείων της ουσών ακτινοβολιών. Ε, γίνονται, ο οργανισμός αυτός κάνει κάποιες επίσημες εκθέσεις, ε, οι οποίες, αν σωστά ξέρω, εγκρίνονται από το σύνολο των εμπειρογνωμόνων. Νομίζω ότι αυτές πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη. Ε, θέλω επίσης να επισημάνω πως παρότι η εκτινοβολία που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα από τις κεραίες δεν αφορά το πεδίο εφαρμογής, δεν είναι στο πεδίο της ε, οδηγίας, πρέπει να το κάνουμε σαφές για να μην, έχουμε, να μην νομίσει κάποιος ότι δεν λαμβάνουμε πρόνοια για αυτό το τομέα αλλά απ' την άλλη μεριά έχουμε και στο μυαλό μας ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξει κάποια άλλη νομοθετική πρόταση δεν είναι σε αυτή τη φάση δουλειά δικιά μας. Τέλος, για το πρακτικό μέρος της υπόθεσης. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, θα ανταποκριθούμε πλήρως στην εξαιρετικά καλή διάθεση της εισηγήτριας Είμαστε εδώ ανοιχτοί για κάθε συνεργασία, για κάθε συζήτηση, έχοντας στο μυαλό μας την ισορροπία. Έχοντας στο μυαλό μας ότι ο μαγνητικός τομογράφος σε σχέση με συγκεκριμένο αριθμό ασθενειών δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλη τεχνολογία, το υπογραμμίζω, και αυτό όχι μόνο είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά αλλά όλοι στο περιβάλλον μας είτε στο κοντινότερο είτε στο μακρύτερο έχουμε γιατρούς που ασχολούνται με αυτό και μπορούν και αυτοί να μας βεβαιώσουν. Ε, από τη μια μεριά λοιπόν να έχουμε αυτό στο μυαλό μας, από την άλλη μεριά να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλοι όσοι εργάζονται σε περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ε, είτε είναι έξω από νοσοκομεία είτε είναι μέσα σε νοσοκομεία πρέπει να απολαμβάνουν της μεγαλύτερης δυνατής επιστημονικά τεκμηριωμένης προστασίας. τα λέω πολύ συγκεκριμένα και τα δύο ζητήματα και τις δύο πτυχές γιατί θεωρώ ότι το μεγάλο ζητούμενο για να μπορέσει η οδηγία να εφαρμοστεί είναι να βρεθεί αυτή η ισορροπία αυτή η χρυσή τομή. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε χρήσιμοι και στους Ευρωπαίους πολίτες που εργάζονται στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και στους Ευρωπαίους πολίτες που χρειάζονται στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για να είναι υγιείς. Σας ευχαριστώ και είμαι πολύ αισιόδοξη για την πορεία της δουλειάς μας και για το αποτέλεσμα. Ε, και Lynn και, και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Σαρτιέ για την εξαιρετική έκθεση. Ευχαριστώ και την Κομισιόν για τη δική τους δουλειά. Εγώ ήμουν εδώ το 2004 όταν θεσπίστηκε η αρχική οδηγία για τις ηλεκτρομανικές ακτινοβολίες και χαίρομαι ότι τόσο οι σοσιαλιστές όσο και το ΕΛΚ άλλαξαν, προχώρησαν σε σχέση με τα τότε αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων και την αξία των τομογράφων. Το θέμα μας έχει ταλαιπωρήσει. Προσπαθήσαμε να πείσουμε συναδέλφου να μην αντικρούσουν την πρόταση της Επιτροπής, η οποία τελικώς εγκρίθηκε. Έχω δουλέψει τότε με τον Επιτροπό Σπίτλα, καθώς και με την ιατρική κοινότητα, για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα του 2004 και ευτυχώ η ιατρική κοινότητα πίεσε και αυτή την Κομισιόν για να πετύχουμε το περίφημο moratorium. Χωρίς αυτό, έχει δίκιο η κυρία Σαρτιέ, Κάποιοι από τους ανθρώπους που ωφελήθηκαν από την μαγνητική τομογραφία θα ήταν σήμερα νεκροί. Ας μην ξεχνούμε λοιπόν ότι μιλάμε για αξιονικούς τομογράφους, τελευταίες τεχνολογίες που βοηθούν τους ασθενείς, αλλά και αυτούς που τους χειρίζονται. Ο σχεδιασμός των τομογράφων καλύτερα από οδηγίες που αφορούν τον ιατρικό εξοπλισμό και από άλλα κείμενα. Υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες για τις συγκεκριμένε συσκευές καθώς και για τους χειριστές τους. Οι διαδικασίες στα νοσοκομεία, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η εκπαίδευση των ε, χειριστών είναι τέτοια που προστατεύουν τους εργαζόμενους. Άλλωστε κανείς από εμά δεν θέλει να διακινδυνεύσουμε την υγεία των εργαζομένων. πριν το 2004 αλλά και μετά. Μίλησα με πολλούς ειδικού και μάλιστα ειδικού που δουλεύουν σε αυτόν τον τομέα και κανείς δεν είπε συμπεριλαμβανομένων των χειριστών επαναλαμβάνω ότι θέλουν να περιορίσουν την χρήση των τομογράφων. Ίσα ίσα οι άνθρωποι αυτοί είναι εκπαιδευμένοι και οι ίδιοι υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να παρέχει αντίστοιχη προστασία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν αυτή τη φορά να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε γιατί εδώ πρόκειται στην κυριολεξία για διλήμματα ζωής ή θανάτου. Κύριε Σαρτιέ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνατε εν ώψη της ε, ενσωμάτωσης της οδηγίας του 2012, ότι είναι να κάνουμε, ας το κάνουμε σήμερα. Έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας και μπορούμε να εξαιρέσουμε τους αξονικούς τομογράφους. Δεν λέω ότι θα εξαιρεθούν οι εργαζόμενοι χειριστές των αξιονικών τομογράφων, όμως οι οριακές τιμές δεν πρέπει να ισχύσουν για τους αξιονικούς τομογράφους. Από εκεί πέρα θα προστατεύσουμε φυσικά και τους χειριστές τους. χειριστές εμπίπτουν στο αντικείμενο, στο πεδίο εφαρμογή της οδηγία. Φυσικά εδώ δεν μιλάμε μόνο για αξιονικούς τομογράφους, μιλάμε και για πολλά άλλα θέματα. Η κυρία Ράπτη έχει δίκιο για τις βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις. Δεν μπορούμε, έχετε δίκιο, να αξιολογήσουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Ίσως να μπορέσουμε να το πράξουμε στο μέλλον. Όμως για τη συγκεκριμένη οδηγία, όπως γνωρίζουμε και από τους επιστήμονες και τις σχετικές έρευνες, δεν μπορούν να αξιολογηθούν. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες στον τομέα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω να μην υπάρχουν κεραίες κινητή τηλεφωνία κοντά στα σχολεία, για παράδειγμα, ή σε παιδικού σταθμού. Όμω για τι μακροπρόθεσμε επιπτώσει ακόμα δεν υπάρχει συνένεση τη επιστημονική κοινότητα. Συνεπώ δεν μπορούμε να ενσωματώσουμε εδώ διατάξει, όπω είπε και η κυρία Ράπτη, οι οποίε δεν θα στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Α μιλήσουμε λοιπόν για τι βραχυπρόθεσμε επιπτώσει. Έχουμε σειρά τροπολογιών. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές τώρα, γιατί το κείμενο της Κομισιόν είναι πολύ καλό. Έχουμε τροπολογίες και από την κυρία Σαρτιέ. Έχουμε όμως συγκεκριμένα την 5, η οποία προβληματίζει ως προς το εξή, γιατί λέει ότι για να παρασχεθεί επαρκής προστασία προς εργαζομένους οι οποίοι δουλεύουν στην γειτονία πλησίων. Τι σημαίνει αυτό, πλησίων. Ε, γιατί χρήζει διαφορετικών, επιδέχεται διαφορετικών ερμηνεών. Επίσης για την απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού και τα σχετικά μηχανήματα όταν λειτουργούν. Τι σημαίνει αυτό. Γιατί, ξέρετε, η αξονική τομογράφη είναι σε λειτουργία ακόμη και όταν δεν καναλούμε έναν ασθενή. Δηλαδή υπάρχουν μαγνητικά πεδία ακόμη και όταν δεν υπάρχει ασθενής μέσα στον εξονικό τομογράφο. Να διευκρινίσουμε λοιπόν περί τίνος πρόκειται εδώ. Να διευκρινίσουμε με άλλα λόγια ότι το μηχάνημα λειτουργεί ακόμη και όταν δεν υπάρχει ασθενής εντός του τομογράφου. Και επίση υπάρχει εδώ άλλη μία τροπολογία που λέει μόνο οι οποίοι επιτρέπεται να είναι πλησίων, του εξοπλισμού κλπ. Τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει επίση. Ε, διενεργούν ιατρικά καθήκοντα. Μην ξεχνάτε ότι τα μηχανήματα αυτά συντηρούνται, καθαρίζονται, με αποτέλεσμα να εκτίθενται και άλλοι άνθρωποι σε ακτινοβολία. Κύριε Σαρτιέ και κύριε Ράπτη, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε στο άρθρο 2 να ξαναδούμε αυτήν την τροπολογία για να διευκρινίσουμε ακριβώ τι σημαίνει το κείμενο. Και υπάρχει και κάτι άλλο στο 4-5 γάμα τροπολογία 6 Αντιλαμβάνομαι τι λέει εδώ το κείμενο για εγγύους και ανθρώπους με βηματοδότες. Εδώ ο εργοδότης για λόγου προσωπικών δεδομένων, προστασία προσωπικών δεδομένων, δεν έχει το δικαίωμα πολλέ φορέ να ρωτήσει και να γνωρίζει εάν μια γυναίκα είναι έγκυο ή αν κάποιο φέρει βηματοδότη. Και για λόγου βεβαίω ισοτιμή μεταχείριση. Το κείμενο τη Κομισιόν προϋποθέτει ότι κάποιος έχει δηλώσει ότι είναι έγκυος ή ότι φέρει το οποίο όμω αντιβαίνει με την νομοθεσία περί ισορροπή μεταχείρισης κλπ. ή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Να το ξαναδούμε λοιπόν και αυτό. Και 5.1. Εκεί έχουμε την τροπολογία υπαριθμών 9. Η τροπολογία η επόμενη επίση αναφέρεται τι έμεσε πιθανέ επιπτώσει από έκθεση. Και εδώ πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό. Δεν λέω ότι διαφωνώ, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λέει το κείμενο. Στο άρθρο 6 έχουμε επίση τα θέματα εκπαίδευση. και οι έμεσε επιπτώσει από την έκθεση. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει ακριβώ. Ποιε είναι οι έμεσε επιπτώσει από την έκθεση. Τι εννοείται εδώ λοιπόν, να το δούμε και αυτό. Άρθρο 8, τροπολογία 12. Σύμφωνο ότι η εξέταση πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Έχω θέμα και με το κείμενο της Κομισιόν εδώ. Εσείς έχετε δίκιο προς την τροπολογία σας. Το κείμενο της Κομισιόν όμως θέλει ακόμη ένα κοίταγμα. Ίσως να πρέπει να το επαναδιατυπώσουμε. Το αρχικό κείμενο παραλαμβάνω της Κομισιόν. Θα βρούμε και με τη δική σας σύμφωνη γνώμη μια νέα διατύπωση. Αυτές ήταν ε, οι σκέψεις μου όσον αφορά συγκεκριμένες πτυχές του κειμένου. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια όμως. Συγχαρητήρια και στην κυρία Ράπτη για τη δουλειά που έκανε επί του θέματος γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι μέσα σε μια γενικότερη κακοφωνία προσπάθησε να προστατεύσουμε τον χώρο των αξιονικών τομογράφων. Λοιπόν, είμαστε όλοι στο ίδιο μήκο κύματο. Ο στόχο είναι κοινό. Ε, πιστεύω ότι θέλουμε να προστατεύσουμε τη δουλειά που γίνεται με του αξιονικού τομογράφου. Και εντελεί και μετά ο λόγο των Κομισιόν, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο που θέλει το λόγο. Η κυρία Ντελή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Ευχαριστούμε την ε, κυρία Μωράν Σαρτιέ για τη δουλειά της. Ε, σας συγχαίρω για αυτήν. Έχω μια σειρά από παρατηρήσεις. Καταρχήν, μόλις εγκρίναμε μια έκθεση, τη δική μου, που ονομάζεται «Ασφάλεια και υγεία στην εργασία». Θεωρώ ότι η, πρωτο, η προτεραιότητα πρέπει να βρίσκεται εδώ σε αυτή την έκθεση και ως εκ τούτου γίνεται με ανεπαρκή τρόπο. Οι εξαιρέσεις γίνονται κανόνας, οι οριακές τιμές καθορίζονται χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση και προχωρούμε περισσότερο προς την κατεύθυνση που προτείνει το Συμβούλιο. Εγώ ε, προτείνω να επανέλθουμε στις τιμές του διεθνούς οργανισμού όπως και για τις ε, βασικές συχνότητες. Η οδηγία θα πρέπει να ισχύσει και για τον τομέα της ε, ιατρικής μηχανικής. Έχουμε τιμές που πάλι έχει ε, δώσει ο Διεθνής Οργανισμός πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας τα συμφέροντα των ε, ασθενών και των εργαζομένων χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο την τεχνολογία. Αλλά αυτοί που λένε το αντίθετο δεν στηρίζονται επιστημονικά. Θεωρούμε ότι οι προτάσεις της εισηγήτριας στην τροπολογία υπαριθμών 5 να αφήσει μόνο στους ίδιους τους εργαζόμενους τον καθορισμό των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που τους ε, ε, αφορούν είναι ανεπαρκής. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες για να εξασφαλιστεί ίση προστασία όλων των εργαζομένων αλλά και για τους κατασκευαστές ώστε να υπάρξει ε, νομική ασφάλεια για τα πρότυπα. Θεωρώ λοιπόν εγώ και το νέο εκ μέρους της ομάδας μου ότι θα θέλαμε να γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων όχι μόνο μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα και ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και να ε, συμπεριληφθεί στο κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. εκπροσωπείται εδώ και η Προεδρία του Συμβουλίου. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν στην Προεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ευτυχής που διαπιστώνει ότι οι περισσότεροι από τους ε, ομιλήσαντες ικανοποιούνται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά τους μαγνητικούς τομογράφους. Όπως είπατε και εσείς, αυτό αποτελεί αποτέλεσμα διαβουλεύσεων που έγιναν ε, με μεγάλη συχνότητα και στις οποίες συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι για να εξασφαλιστεί ένας καλός συνδυασμό ανάμεσα στην αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και τη δυνατότητα λειτουργίας και ανάπτυξη αυτών των συσκευών. Ε, συμφωνούμε όλοι ότι η χρήση των ε, της μαγνητικής ε, απεικόνησης είναι απαραίτητη. Επίσης βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύμανος με πολλούς από τους ομιλητές όσον αφορά την επιστημονική επάρκεια που χρειάζεται για να δικαιολογηθούν για να παρακολουθηθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όμως ε, και η Κομισιόν θα παρακολουθήσει. Παρά τα αυτά, η κυρία Ράπτη είπε κάτι. Οι τηλεφωνικές κεραίες, όταν πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν συντήρηση στις κεραίες αυτές, καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Δηλαδή το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας καλύπτει όλους τους εργαζομένους παρότι για κάποιες κατηγορίες υπάρχουν μικρές διαφορές όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Επίσης, η κυρία Ντάλη είπε ότι θα προτιμούσε την επιλογή του Συμβουλίου. Εγώ επιμένω, τα προσαρτήματα 2 και 3 της πρώτης Κομισιόν στηρίζονται και αυτά ακριβώς σε αυτές τις τιμές του Διεθνούς Οργανισμού, της Διεθνούς Επιτροπής. Αυτές ακριβώς δημοσιεύθηκαν τον Νοέμβριο του 2010 για τις χαμηλές συχνότητες. Ήταν πολύ αργά και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να δείξουμε τα αποτελε... τη... Το... Το... δουλειά μας νωρίτερα και παρουσιάζονται με τέτοιο... τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί και η προστασία των εργαζομένων αλλά και η λειτουργία των περισσότερων δραστηριοτήτων με τρόπο συνεκτικό και αποτελεσματικό. Επιμένω, η Κομισιόν τήρησε τις και τις τιμές ε, του Διεθνούς Οργανισμού. Και για να επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η κυρία Λίν, πράγματι στην τροπολογία επαριθμών 5 θα πρέπει ίσως να αλλάξουν κάποια, κάποιες λεπτομέρειες γιατί πράγματι προβλέπεται δύο τρόποι λειτουργίας των συσκευών όταν είναι stand-by ή όταν ε, υπάρχει στατικό ηλεκτρο, ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ή όταν γίνεται η, ε, η ιατρική εξέταση ή η δοκιμή της συντήρησης όπου υπάρχουν υψηλές συχνότητες, πεδία υψηλών συχνοτήτων. Πρέπει να γίνει η διάκριση γιατί ένας ε, μαγνητικός τομογράφος δεν είναι συσκευή που ανάβει και κλείνει με έναν διακόπτη ή χρειάζονται μέρες για να αποκατασταθεί η σταθερότητά του. Αυτά με δύο λόγια. Ε, ήθελα να πω από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ το Κοινοβούλιο που έκανε δεκτή την πρόταση αυτή η οποία πρέπει να πω ότι δεν έγινε στο πόδι. Ε, πραγματικά επιδιώξαμε να έρθουμε σε επαφή και να ακούσουμε στις ομάδες εργασίας όλους όσοι το επιθυμούσαν για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Μοχον Σοντιέ, για όλα αυτά τα οποία έχει προσφέρει μέχρι σήμερα. Είχαμε πάρα πολλές συζητήσεις για το θέμα αυτό. Η Πολωνική Προεδρία εργάστηκε πολύ σκληρά για να καταλήξει στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε ομάδα εργασίας και ομάδε εμπειρογνωμόνων. Ε, σε πέντε μήνες λοιπόν σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο και ε, αυτό το, την τελική μας σύγηση θα την καταθέσουμε στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Όσον αφορά τώρα το κείμενο της οδηγίας, επ' αυτού σε μεγάλο βαθμό υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν βέβαια δύο θέματα που εκκρεμούν ακόμα και πρέπει να στηθούν. Είναι το παράρτημα υπαριθμών 2 για τις οριακές τιμές και κατόπιν υπάρχει και το θέμα της ε, διατύπωσης για τις εξαιρέσεις. Για αυτά τα δύο θέματα το Συμβούλιο θα συνεχίσει την εργασία του. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει πλήρης ε, σαφήνεια και εγώ ε, θα ήθελα να συμπληρώσω αυτά που είπε η συγγήτρια αναφέροντας τα εξής. Η συγγήτρια είπε ότι η Πολωνία είναι μία από τις χώρες ε, που μπλοκάρει το θέμα των εξαιρέσεων. Αλλά ξέρετε η Πολωνική Προεδρία αποφάσισε να μην παραμείνει άκαμπτη σε κανένα θέμα της οδηγίας με τον τρόπο αυτό να ανοίξει τον δρόμο για συμβιβασμό. Έτσι λοιπόν η δική μας η θέση είναι αμερόληπτη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε τελική ανάλυση δεν θα τοποθετηθούμε και εμείς. Ευχαριστώ. Η κυρία Σιγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους που είναι ε, συντάκτες από τις ε, άλλες πολιτικές ομάδες όπως επίσης τους εκπροσώπους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Σημείωσα όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν. Επιμένω σε αυτό που είπε η κυρία Λίν ότι οι, οι τομογράφοι ε, καλύπτονται ήδη από οδηγία και ότι εδώ και πολλά χρόνια όλη η πρόοδος που σημειώθηκε στην κατασκευή αυτών των συσκευών ε, προσπαθεί να περιορίσει την έκταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου ώστε ε, να προστατεύεται και η υγεία των ασθενών και των εργαζομένων, αλλά τα ίδια ίδιες οι συσκευές προστατεύονται, έχουν συστήματα προστασίας και αυτοί οι οποίοι εργάζονται με αυτά ε, βρίσκονται σε χώρο ε, χωριστό από αυτό των μηχανημάτων εκτός από κάποιες πολύ συγκεκριμένες και σπάνιες περιπτώσεις ε, παραδείγματο χάρη όταν εμπλέκονται παιδιά. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να επιμείνω είναι ότι χαίρομαι πολύ που διαστάνουμε ότι υπάρχει μια συνολική θέληση, μια σύγκληση στην επιθυμία να επιτύχουμε, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι αν δεν καταφέρουμε να περάσουμε μια τέτοιου είδους οδηγία με στόχους τους οποίους συμμεριζόμαστε όλοι, το 20% σχεδόν των ασθενών θα στερηθούν από μια σειρά, μια εξετάσεων ε, τα άτομα με αναπηρία, τα παιδιά κτλ. Και βεβαίως ε, θα υπάρξει ένα σημαντικό κενό ε, για την υγεία των συμπολιτών μας, για μας τους ίδιους ίσως αύριο. Το τρίτο θέμα είναι το εξής. Υπάρχουν πάρα πολύ καλογραμμένοι οδηγοί χρήσης που μπορούμε να αναφέρουμε και συγκεκριμένα και που μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για να διευκολυνθεί η προστασία των εργαζομένων. Εν πάση περιπτώσει, ναι, κύριε Λίν, πρέπει να είναι καθαρό το αντίγραφό μας. Ναι, κύριε Ράπτη, πρέπει να δουλέψουμε με βάση επιστημονικά στοιχεία και να μην ε, ε, δημιουργηθούν προβλήματα από ανύπαρκτες δυσκολίες. Θέλω επίσης να πω στην Μαντελή ότι για το θέμα που έθεσε. Πράγματι, όπως είπε ο κύριος Ερμπιγιόν, οι τιμές της Διεθνούς Επιτροπής έχουν ληφθεί υπόψη στους πίνακες των τιμών ορίου των οριακών τιμών. Άρα το αίτημά σου Καριμά έχει ήδη ληφθεί υπόψη στο κίνημα. Μην κάνουμε λάθος σε αυτή την περίπτωση ενώ από την άλλη πλευρά η προστασία των εργαζομένων στον ιατρικό χώρο και στις ιατρικές δραστηριότητε, είτε πρόκειται για συντήρηση είτε καθαρισμό των χώρων αυτών φυσικά είναι κάτι που πρέπει να καλυφθεί. Τέλος, πιστεύω ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να προχωρήσει θετικά και επ' αυτού του θέματος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να υπάρξει υπερβολική διάσταση μεταξύ της δουλειάς του ενός και του άλλου που, πράγμα που θα καθυστερήσει την οδηγία αυτή που περιμένουμε. Τέλος θα ήθελα να σας πω ότι σημείωσα τις παρατηρήσεις ε, για τις ε, προβληματικές τροπολογίες. Είμαι στη διάθεσή σας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά. Οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε υποχρέωση να είμαστε αποτελεσματικοί και ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε διότι είναι μια δουλειά προσφυλή σε όλους μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ. Όπως είπατε, οι τροπολογίες μπορούν να καταρριφθούν μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. 25 ε, Ιανουαρίου θα τις εξετάσουμε και θα ψηφίσουμε κατά τη διάρκεια έκτακτη συνόδου της Επιτροπής μας. 13 Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο κατά το οποίο σημαίνει ότι είναι αρκετά λογικό το χρονοδιάγραμμα και συμβατώ με αυτό του Συμβουλίου. Οπότε κλείσαμε με το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης και μπορούμε να περάσουμε στο υπαριθμό 16 παρουσίαση από την Επιτροπή των προτάσεων για την τροποποίηση του κανονισμού που αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ο κ. Λεμπρά είναι εδώ εκ μέρου τη Κομισιόν. Βεβαίω, στην ομάδα εργασία τη Επιτροπή ΦΕΜ ε, ακούσαμε 18 Οκτωβρίου και 9 Νοεμβρίου αντίστοιχε παρουσιάσει, όμω δεδομένου ότι το κείμενο είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Επιτροπή μα γενικώ, ε, έκρινα χρήσιμο και μάλιστα απαραίτητο να συζητήσουμε το θέμα ακριβώς αυτό. Κύριε Λεμπρά, παρακαλώ έχετε τον λόγο για να μας παρουσιάσετε τις προτάσεις της Κομισιόν. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Συνοδεύομαι από δύο συναδέλφους της Γενικής Διεύθυνσης ε, Γεωργίας, Άγκρη, στην περίπτωση που τεθούν ερωτήματα σχετικά με την επέκταση του Ταμείου στους αγρότες. Επενθυμίσω καταρχήν την υφιστάμενη κατάσταση, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των προτινομένων τροποποιήσεων. Το EGF, το, Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαμωγής στην Παγκοσμιοποίηση, παρεμβαίνει στις περιπτώσεις μαζικών απολύσεων που προκαλούν προβλήματα που έχουν σχέση με την παγκοσμιοποίηση αλλά και στην περίπτωση προβλημάτων που έχουν σχέση με την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση για μια συγκεκριμένη περίοδο, μια πεπερασμένη περίοδο, ως τα τέλη της χρονιάς δηλαδή. Εμείς προτείνουμε επέκταση αυτή αυτής της χρονικής περίοδου. Θα παραλέψω σε αυτό κυρία Πρόεδρε. Παρεμβαίνουμε μόνο στις περιπτώσεις μαζικών απολύσεων. με ελάχιστο κατώτερο όριο του 500 εργαζόμενους για περίοδο 4 έως 9 μηνών. Υπάρχει δηλαδή συγκέντρωση και στο χρόνο και στο αντικείμενο. Προσφέρουμε στους εργαζόμενους. Συγχρηματοδοτούμε δηλαδή, αν θέλετε, μέσω του Ταμείου ένεργα μέτρα παρέμβαση στην αγορά, δηλαδή η εκπαίδευση, η παροχή συμβουλών, κατάρτιση, επιχειρηματικότητας κλπ. Υποστηρίζουμε επίση το εισόδημα κατά τη διάρκεια λήψη και υλοποίηση αυτών των μέτρων. Και αυτό για 24 μήνες το πολύ, με συγχρηματοδότηση που ανέρχεται σε 50% του συνόλου, ποσοστό το οποίο ανέρχεται πλέον σε 65% κατά την περίοδο της εξαίρεσης λόγω κρίσης. Προπολογισμός 250 εκατομμύρια. Να μην ε, αναφερθώ και πάλι στα γνωστά, υπενθυμίζω απλώς ότι έχουμε καλύψει ως τώρα 76.000 εργαζόμενους στην Ευρώπη για συνολικό ποσό 350 εκατομμύρια ευρώ. 70 εκατομμύρια κατά μέσο το χρόνο. Στα δύο τρίτα των περιπτώσεων ενεργοποιείται η εξαίρεση λόγω κρίσης. Δηλαδή, σε 20 περιπτώσεις μόνο, 4 με 5 περιπτώσεις μόνο το χρόνο αφορούν μόνο αποκλειστικά την παγκοσμιοποίηση. Θα παρέλθω στην αξιολόγηση του Ταμείου προς το τέλος και συνεχίζω λέγοντας ότι αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να υποβάλει νέα πρόταση για την περίοδο 2014-2020 η οποία θα βασίζεται στην λεγόμενη προσθεμένη αξία του Ταμείου. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν και πάλι μαζικές απολύσεις, ανεξαρτήτως του αν ε, συμβαίνουν σε ένα συγκεκριμένο χώρο, σε μια ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε να είμαστε σε θέση να παράσχουμε πιο αποτελεσματική ενίσχυση να συγχρηματοδοτήσουμε και προγράμματα του κοινωνικού ταμείου προσαρμοσμένα και στις ατομικές ανάγκες για μεγαλύτερες περιόδους. Εδώ εμπλέκουμε και τους κοινωνικούς εταίρους σε διάφορα επίπεδα. όχι μόνο κατά τη διάρκεια των απολύσεων, αλλά και για την εξέβρεση των καταλληλών μέτρων και την υλοποίησή τους. Εμπλέκονται επίσης τοπικοί και περιφερειακοί εταίροι για το σκοπό της υλοποίηση των σχετικών μέτρων. Πρόκειται για αλληλεγγύη, δεν υπάρχει εδώ εθνικό ανατοτόριο συμμετοχής. Το Ταμείο λαμβάνει υπόψη του την επικουρικότητα, γιατί όπως προείπα, συγχρηματοδοτούμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο. Η Κομισιόν προτείνει συναφώς όπως προείπα, να επεκτείνουμε τον ρόλο του Ταμείου για να καλύψουμε και τη γεωργία στην περίπτωση που υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις από μεγάλες εμπορικές συμφωνίες. Τα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, πρόκειται για αντιμετώπιση της κρίσης, συνεπώς δεν προβλέπεται ετήσιον το όριο. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να είχαμε πει 400 εκατομμύρια ευρώ, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσουμε μικρότερα ή υψηλότερα ποσά. Παρότι το όριο, ο συνολικό προπολογισμό είναι 3 δισεκατομμύρια για την τρέχουσα περίοδο. Για την προηγούμενη φάση είχαμε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε λοιπόν μια μικρή μείωση. Υπενθυμίζω όμω ότι ω σήμερα χρησιμοποίησαμε μόνο 350 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια των πρώτων 5 ετών. Όσον αφορά τώρα τους αγρότες, προβλέπουν νέες προτάσεις ότι ένα μέρος του προπολογισμού των 3 δισεκατομμυρίων έως και 2,5 δισεκατομμύρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον τομέα της γεωργίας. Έως και, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το ανώτατο όριο, 2,5-3 δισεκατομμύρια από τα 3. Λίγα λιγότερα από τα προηγούμενα 3,5. Τις αιτήσει υποβάλλουν τα κράτη-μέλη. Η περίοδος αναφοράς 4 έως 9 μηνών παραμένει το κατώτατο όριο των 500 απολύσεων συνεχίζει να ισχύει. Όμως έχουμε πλέον την δυνατότητα να επεμβαίνουμε και σε μικρότερες αγοράς εργασίας ή στην περίπτωση εκτάκτων περιστάσεων όπου ενδεχομένως το κατοχληστό των 500 εργαζομένων δεν μπορεί να τηρηθεί λόγω του ότι πρόκειται για μια πολύ μικρή χώρα ή στην περίπτωση που παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλες απολύσεις, οι απολύσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα μια τοπική σημαντική κρίση. Το κατόφλι, το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης παραμένει 50%. Ο σκοπός μας είναι να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο την χρηματοοικονομική κρίση, αλλά και οποιασδήποτε άλλες κρίσεις σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε ένας μόνιμος μηχανισμός, ο οποίος ε, θα προσφεύγει στους πόρους του Ταμείου. Στις περιπτώσεις, για παράδειγμα, απρόσμενων τοπικών κρίσεων, εκεί το EGF, το Ταμείο, θα μπορεί να παρεμβαίνει. Και όχι μόνο αυστηρά στις περιπτώσεις επιπτώσεων από την παγκοσμιοποίηση. Επίσης, οι επισυμβάσει, οι υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίε, οι εποχικοί εργαζόμενοι, οι μικροί ανεξάρτητοι επαγγελματίε και αυτοί θα μπορούν πλέον να μπορούν να αποφελούνται από το Ταμείο και όχι μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι. Εστιάζουμε ακόμη περισσότερο τη δράση μας στα ενεργά μέτρα στην αγορά εργασίας. Για τα μέτρα αυτά κρατάμε κατελάχιστον έναν προπολογισμό 50% της παρέμβασής μας. Το ποσοστό της χρηματοδότησης όμως του EGF αυξάνεται όπως είπα σε 65% στην περίπτωση ιδιαίτερα δύσκολων κρίσεων σε περιφερειακό επίπεδο σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Έχουμε όμως και άλλες βελτιώσεις. Μπορούμε να καλύψουμε πάνω από δύο περιφέρειες ταυτόχρονα. αντιμετωπίσαμε κρίσεις όπως η ε, τυπογραφία στις ε, κατοχώρες. Σε άλλες περιπτώσεις ε, είχαμε αιτήματα τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν να καλύπτουν για παράδειγμα ακόμα και όλη την επικράτεια μιας χώρας όπως προκειμένου της Ολλανδίας. Μπορούμε πλέον λοιπόν να καλύπτουμε πάνω από μία περιφέρεια. Υπάρχει συνεπώς μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση των μέτρων. Τα μέτρα θα είναι πιο εύκολο να τροποποιηθούν και τούτο γιατί διαπιστώσαμε κάποιες ακαμψίες στο παρελθόν που δεν μας επέτρεπαν να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κατάρτισης ή τις συγκεκριμένε ανάγκες κάποιες περιοχής. Επίσης, η διαδικασία υποβολής αίτησης θα απλουστευτεί για να μπορούμε να παρεμβαίνουμε και πιο γρήγορα. Η ανάλυση επίσης της εκάστοτε αίτησης θα γίνεται πιο γρήγορα. Υπάρχει ένα ανώτατο όριο ε, εβδομάδων τόσο για την Κομισιόν όσο και για το κράτος μέλος για να μην επανεληφθούν κάποια φαινόμενα της προηγουμένης περίοδου όπου χρειάστηκε ε, περιμένουμε μήνες έως και πάνω από ένα χρόνο από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης έως την επεξεργασία και την λήψη της τελικής δημοσιονομικής απόφασης λόγω ακριβώ των ε, μακροχρόνων συνομιλιών με το κράτος μέλος. Επίσης, θέσαμε έναν στόχο την επανένταξη του 50% τουλάχιστον των εργαζομένων με την έννοια ότι αυτός ο στόχος είναι ένας έλεγχος της απόδοσης των μέτρων μας θα είναι μια απόδειξη δηλαδή, ότι τα μέτρα ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες. Κάτι νέο εμπροκειμένο πολύ σημαντικό κατά τα άλλα είναι η συμπερίληψη των αγροτών, οι οποίοι θίγονται από τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ η μόνη διαφορά είναι ότι ο μηχανισμός ενεργοποίησης του Ταμείου είναι λίγο διαφορετικός. Για τα άλλα μέτρα παραμένουμε στο γνωστό υφιστάμενο πλαίσιο. θα διερωτηθεί κάποιος γιατί οι αγρότες. Πρώτον, γιατί οφείλουμε να καλύψουμε όλους τους τομείς και δεύτερον, διότι οι συμφωνίες ε, Mercosur είτε η ατζέντα της Ντόχα ε, είναι συμφωνίες οι οποίες έχουν μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Εμεί κάτι πρέπει να κάνουμε για τι αρνητικέ επιπτώσει αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του Μερκοσούρ ξέρουμε ότι η Γεωργία θα μπορούσε να χάσει έω και 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω ακριβώ των συμφωνιών Μερκοσούρ. Ο τομέα βεβαίως γενικότερα τη βιομηχανία θα μπορούσε να κερδίσει 8 δισεκατομμύρια από αυτή την υπόθεση και ο τομέα των υπηρεσιών περίπου 17 δισεκατομμύρια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λοιπόν λογικό, έχοντα αυτά τα ωφέλη από τη μία πλευρά, να παρεύουμε στην άλλη μέσω του Ταμείου και να κάνουμε κάτι για αυτούς που έχουν να χάσουν από τέτοιες συμφωνίες. Είναι αν θέλετε μια μεταφορά από τους κερδισμένους ούτως υπήν προς τους χαμένους αυτών των εμπορικών συμφωνιών. Όπως προείπα, αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κατάλληλου μηχανισμού με βάση την εξή διαπίστωση. Οφείλουμε να διατηρήσουμε έναν γεωργικό πληθυσμό στην Ήπεθρο και μάλιστα έναν πληθυσμό ο οποίος θα έχει δραστηριότητες και αντικείμενο. Γι' αυτό ακριβώ πρέπει να είμαστε σε θέση να παρεμβαίνουμε πριν την οριστική πάυση της γεωργικής δραστηριότητας. Πρέπει επίσης να είμαστε σε θέση να προβλέπουμε τις αρνητικές επιπτώσεις. Προς τον σκοπό αυτό, η Κομισιόν με βάση τις εκ των προτέρων αναλύσεις της, αλλά και βάση των παρατηρήσεων, των τιμών, των προϊόντων, των εισαγών κλπ. Η Κομισιόν λοιπόν, επαναλαμβάνω, θα προτείνει για σειρά προϊόντων τα οποία θίγονται κατά τη διάρκεια της περίοδου αναφοράς και με βάση συγκεκριμένε προποθέσει, Η Κομισιόν λοιπόν θα προτείνει στα κράτη-μέλη να υποβάλουν αιτήσει για τους στιγόμενου αγρότες. Φυσικά το κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τις πραγματικές αρνητικές επιπτώσει επί των αγροτών πριν υποβάλει την σχετική αίτηση. Ενώ λοιπόν ότι από μια μεριά έχουμε τα γενικά στατιστικά στοιχεία, παράλληλα όμω πρέπει να συντρέχουν και άλλοι λόγοι, οι συγκεκριμένε περιστάσει δηλαδή, σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή. Το EGF επίσης μετά από 15 μήνε θα υποβάλει την προσωρινή, την ενδιάμεση έκθεσή του, αυτό είναι μία από τι νέε προτάσει, Και ένα άλλο νέο, μια νέα διάταξη αφορά την ανάγκη και τον στόχο επανένταξη στην αγορά εργασία τουλάχιστον των 50% των απολυμμένων εντό περίοδου 12 μηνών. Εδώ μα ενδιαφέρει προσπάθεια, όχι τόσο το απόλυτο νούμερο. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν συγκεκριμένε προσπάθειε σε συγκεκριμένε περιοχέ, οι οποίε να επικεντρώνονται περισσότερο σε αυτόν τον στόχο σε σχέση με άλλε περιοχέ. Το κράτο μέλο δηλαδή πρέπει να θεσπίσει μέτρα με στόχο την ε, αντιμετώπιση των δυσκολιών που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι στην επανένταξή του στην αγορά εργασία. Και επανέρχομαι τώρα στι συστάσεις που προέκυψαν από την ενδιάμεση έκθεση. Να ανοίξω όμως πρώτα μια παρένθεση θα δώσω στη γραμματεία σας την Δευτέρα ή την Τρίτη την περίληψη και τις πολιτικές συστάσεις που προέκυψαν από την ενδιάμεση αξιολόγηση. Το πλήρες κείμενο της έκθεσης θα είναι διαθέσιμο περί τα μέσα Δεκεμβρίου. Όμως έχουμε ήδη στη διάθεσή μας και πολύ γρήγορα θα έλεγα την περίληψη και τις συστάσεις πολιτικής. Γιατί επιταχύνουμε αυτήν την διαδικασία. Αυτό συνδέεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε αυτή τη ε, στιγμή στο Συμβούλιο σχετικά αφορά την εξέρεξη λόγω κρίσης. Στις 2 Φεβρουαρίου θα διοργανωθεί μια ευρεία σύσκεψη με άλλους εμπλεκόμενους και κοινωνικούς φορείς για να συζητήσουμε ακριβώς την ε, ενδιάμεση αξιολόγηση. Όμως μπορώ ήδη από σήμερα να σας πω ως προς τις ε, συστάσεις τα εξής. αντιμετωπίσουμε αίτημα μείωση του αρχικού κατοφυλίου των χιλίων απολυμμένων, το αρχικό όριο. Αυτό το πράξαμε από το 2009, το όριο αυτό κατέβηκε στους 500 απολυμμένους. Μάλιστα το όριο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τρόπο πιο ευέλικτο και δει σε έκτακτες περιπτώσεις ή σε μικρές αγορές εργασίας. Έτσι μπορούμε να ικανοποιήσουμε επιπλέον αιτήματα. Επίσης ικανοποίησαμε το αίτημα συμπερίληψης και των επισυμβάσεων εργαζομένων. Από την άλλη μεριά διατηρήσαμε τη διάρκεια της περίοδου αναφοράς κάπου μεταξύ 4 και 9 μηνών εντός των οποίων πρέπει να γίνει και η μαζική απόλυση. Όσον αφορά την εφαρμογή του μέτρου μας ζήτησαν επίσης να παρατείνουμε την περίοδο υλοποίηση των μέτρων. Και όντως από 12 μεγαλώσαμε αυτήν την περίοδο σε 24 μήνες. Όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, ζητήθηκε επίσης η παρακολούθηση αυτή να αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης και αυτό θα γίνει με την έκθεση που θα υποβληθεί 15 μήνες αργότερα. Ζητήθηκε επίσης πιο αποτελεσματική ανταλλαγή καλών πρακτικών. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε περισσότερη τεχνική βοήθεια έτσι ώστε το EGF, το Ταμείο, να είναι και πιο ορατό, η δράση του να γίνει πιο αισθητή. Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την εξαίρεση λόγω κρίσης, να πω δύο λόγια για την κατάσταση στο Συμβούλιο. Στις 10 Ιουνίου υποβάλαμε πρόταση για την παράταση της εξαίρεσης για τα δύο τρέχοντα έτη, 2012-2013 ε, δηλαδή, με την έννοια ότι κανονικά η εξαίρεση αυτή θα έπαβε στις 31 Δεκεμβρίου του 2011. Προτείναμε επίσης να αυξήσουμε το ποσοστό συγχρηματοδότηση στο 65%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε στις 29 Σεπτεμβρίου με την πρότασή μας. Στο Συμβούλιο έγιναν τέσσερις συσκέψεις της ομάδας κοινωνικών θεμάτων. Συνδέησε δύο φορές η Κορεπέρ και δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν κατέστη δυνατόν το Συμβούλιο να καταλήξει σε κοινή θέση. Έξι κρατημέλη, μία, μία ψηφία έχει μπλοκάρει το θέμα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εάν το Συμβούλιο δεν μπορέσει να βρει συμβαστική λύση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2011 επανερχόμεθα στην βασική σχετική νομοθεσία όσον αφορά δηλαδή τις περιπτώσεις ενεργοποίησης του Ταμείου Καταργείται δηλαδή η εξαίρεση και από εδώ και πέρα μόνο θα παρεμβαίνουμε μόνο σε περιπτώσεις, σε περιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση. Το αποτέλεσμα θα είναι να χρησιμοποιήσουμε μόνο το 1 τέταρτο των δυνατοτήτων του Ταμείου από εδώ και πέρα. Η σχετική συζήτηση, η επόμενη σχετική συζήτηση θα γίνει στο Συμβούλιο στην ομάδα κοινωνικών ε, υποθέσεων στο Συμβουλίο την 1η Δεκεμβρίου, όπω ε, είπα. Κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την πρόταση τη Κομισιόν για την νέα μορφή του Ταμείου. Αυτέ είναι οι δυσκολίε όσον αφορά την παράταση τη ισχύω τη εξαίρεση λόγω κρίση. Να θυμίσω μόνο ότι σε λίγε μέρε θα έχετε ε, νέα από εμά την περίληψη και τι προτάσει. Ευχαριστώ. Κύριος Κρότσμαν δεν είναι αλλά έχει εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών. Η κυρία Χάρκιν, η συγγήτρια και μετά η κυρία Κορνίλσεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την παρουσίαση που μας έκανε σήμερα το πρωί. Ήδη στην ομάδα εργασία είχαμε κάποιες πρώτες συζητήσεις. Το πρώτο μου σχόλιο αφορά αυτό που είπατε στο τέλος σχετικά με την εξαίρεση για την κρίση. Αυτό τώρα που θα πω είναι καθαρά προσωπική μου άποψη και το καθιστώ απόλυτα σαφές. Δεν είναι απαραίτητα η άποψη της πολιτικής μου ομάδας. Αλλά πραγματικά σοκάρομαι από το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν αναγνωρίζει την ανάγκη ότι είναι απαραίτητη να υπάρχει κάποια παρέμβαση στο πλαίσιο αυτής της εξαίρεσης. Αν δούμε λιγάκι τα στοιχεία θα διαπιστώσουμε ότι ο αριθμός των αιτήσεων στο πλαίσιο αυτής της εξαίρεσης αυξάνεται κάθε χρόνο από το 2009 και αυτό ήταν αναμενόμενο. Κάθε τρίμηνο παρουσιάζεται μία περαιτέρω αύξηση. Το να κλείνει κανείς τα μάτια του μπροστά σε αυτό, πέρα από το ότι είμαστε στο χείλος του γκρεμού, αυτό δεν νομίζω βέβαια ότι είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει απαραίτητα σήμερα, αλλά δεν καταλαβαίνω ποια, ε, ποιο είναι το πρόβλημά τους. Διότι αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα με το ίδιο το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, αυτό μπορεί να εξεταστεί το πρόβλημα όταν θα εξεταστεί ο νέος κανονισμός. Αλλά αυτή τη στιγμή να μπλοκάρεται αυτή η εξαίρεση για την κρίση, κατά την άποψή μου, είναι απαράδεκτο. Και έτσι λοιπόν, εξετάζοντας ε, και πάλι αυτά που μας είπατε, την ενημέρωσή σας, είπατε όταν υπάρχει διαβούλευση ε, ζήτησαν υπάρξει διαβούλευση 25 κράτη και ε, όλοι συμφώνησαν, οι περισσότεροι συμφώνησαν στο να υπάρχει παρέμβαση όταν υπάρχουν απολύσεις. Δεν ξέρω, είτε οι άνθρωποι να άλλαξαν γνώμη, είτε πέρασε η κρίση, εν πάση περιπτώσει. Ε, θα ήταν πραγματικά πολύ αρνητικό το μήνυμα να πούμε ότι από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους θα πρέπει να επανέλθουμε μόνο σε αυτό το θέμα το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης. Αυτή δεν είναι η προσωπική μου άποψη. Κατά τα άλλα θα κάνω πολύ σύντομα σχόλια γιατί με ενδιαφέρει να ακούσω και τι θα πούν οι συνάδελφοι. Προφανώς λοιπόν συμφωνώ με το ότι οι προσωρινά απασχολούμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, αυτοί μπήκουν στο ταμείο. Ένα σχόλιο που θέλω να κάνω αφορά τα ποσοστά της συγχρηματοδότησης. Άκουσα ότι υπάρχουν ε, ποσοστά συγχρηματοδότησης μέχρι και 25% ε, εγώ δεν ήμουν σε αυτό το ταξίδι στην Ισπανία, αλλά εκεί προέκυψε ένα πολύ χειρό μήνυμα ότι τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο, ή περιοχές, όχι μέλη, περιοχές έχουν δυσκολία να αποκτήσουν πρόσβαση στο ταμείο λόγω ακριβώς των ποσοστών συγχρηματοδότησης και προφανώς ε, προτιμούν το κοινωνικό ταμείο γιατί έχουν μόνο τόσα χρήματα που να μπορούν να προσφέρουν και μερικές φορές ε, για αυτό το λόγο δεν καταφεύγουν στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Εγώ, κατά την άποψή μου, το 65% είναι το ελάχιστο. Ε, ξέρω ότι είχαμε συζητήσει στην Επιστροπή και θα ήθελα επίσης να πω ότι έχουμε και ε, μεταβατικές ε, περιοχές που μόλις έχουν βγει από τη σύγκληση που είναι περίπου στο 78 70 ή 80% και αυτές έχουν το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης που έχουν ΑΕΠ 120-140%. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι και εδώ χρειαζόμαστε ευελιξία. Ίσως αυτό ε, μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω στην Επιτροπή μας. Κατά τα άλλα, η σημαντικότερη αλλαγή Εντάξει, υπάρχουν πολλές αλλαγές, αλλά πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι με την πρόταση περί μεγαλύτερης ευελιξίας, το γεγονός ότι όλη η διαδικασία επιταχύνεται από την ώρα που υποβάλλεται αίτηση μέχρι την τελική της έγκριση, γιατί αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε τη διαδικασία, προφανώς και το στηρίζει η Επιτροπή μας. Πάμε τώρα στους αγρότες. Εκεί διαφωνώ με την Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Εσείς μιλήσατε για μια κατάσταση όπου όλοι είναι ωφελημένοι. Λέτε ότι η Γεωργία, τουλάχιστον έτσι άκουσα, ε, θα πάρει 6,8 δις, η βιομηχανία 8 και οι υπηρεσίες 6,9. Ε, εγώ διαβάζοντας το έγγραφο σχετικά με τη γεωργία και το, τις ενδεχόμενες απώλειες δεν είδα τα στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών και την βιομηχανία. Υποθέτω ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, αλλά ίσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μα δώσει περαιτέρω πληροφορίε από αυτού. Μιλήσατε λοιπόν για την κατάσταση όπου όλοι θα είναι ωφελημένοι, μιλήσατε για την ψυχική ασφάλεια και άλλα θέματα. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί τα 2,5 δις αναφέρονται στον κανονισμό του Ταμείου. Γιατί μιλάμε εδώ για απώλεια, με συγχωρείτε, απώλεια της Γεωργίας κατά 4,8 δις. Και θέλω να ρωτήσω, ε, αυτή η απώλεια για πόσο χρονικό διάστημα υπολογίζεται, για, ποιο, ε, για ποια περίοδο μιλάμε, πόσα χρόνια. Δεν ξέρω βέβαια για άλλα μέλη, αλλά εγώ αυτά τα θέματα με απασχολούν πολύ και ξέρετε ότι πάνω από τα 2,5 δις για τη Γεωργία εμένα μου δημιουργεί πρόβλημα. Φαίνεται ότι τώρα κατά κάποιον τρόπο χρησιμοποιούμε το Ταμείο ως ένα ανάχωμα κατά κάποιον τρόπο για να αντισταθμίσουμε αυτά τα οποία κάνουμε με την εμπορική μας ε, πολιτική. Ε, δεν νομίζω όμως ότι το Ταμείο είχε προβλεφτεί γι' αυτό το σκοπό. Κυρίως αν διαβάσει κανείς τα έγγραφα για το Ταμείο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτό θα ήταν ε, ο στόχος δημιουργίας του. Όπως σας είπα εξετάζουμε τη δυνατότητα των 500 εκατομμυρίων, μισού δις ε, για όλο το χρονικό διάστημα για τους απολυμμένους και εντάξει αυτό χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα το ποσό. Ξέρουμε βέβαια ότι αυξάνονται συνεχώς οι αριθμοί και θα χρειαστεί ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό. Εγώ λοιπόν βρίσκομαι εδώ μεταξύ σκύλα και χάριβδο, αν θέλετε, διότι η άλλη επιτροπή στην οποία είμαι αρμόδια είναι η Γεωργία. Και ανησυχώ ιδιαίτερα για την πρόταση κομισιόν. Εντάξει, θα το κουβεντιάσουμε αλλού αυτό. Εδώ όμω θέλω να πω ότι ένα ταμείο το οποίο υποτίθεται ότι θα προσφέρεται για απολυμμένους εργαζόμενους και αυτή είναι η άποψή μου εγώ δεν έχω πρόβλημα με την πρόσβαση των γεωργών στο ταμείο αυτό όποιος χάνει τη δουλειά του κατά την άποψή μου πράγματι θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο ταμείο αυτό όμως να ξέρουμε ότι η Κομισιόν λέει ότι τα 2,5 δις ε, αυτού του ταμείου θα χρησιμοποιηθούν ως ένα είδος αναχώματος για την απώλεια των 4,8 δις στη Γεωργία, αυτό κατά την άποψή μου εμένα τουλάχιστον δεν με βρίσκει σύμφωνη. Ευχαριστώ. Το λόγο θα δώσω στον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Άγκρη που βρίσκεται εδώ, αλλά αν δεν έχουν αντίρρηση οι συνάδελφοι να το κάνουμε τώρα και ζητώ συγγνώμη την κυρία Χάρκιν θα έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα θα ήταν χρήσιμο, είναι χρήσιμο ε, να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το είδος των διατάξεων που διαμορφώνονται για τους αγρότες είναι διαφορετικά ακόμα και για το ε, σημείο που θα ξεκινήσει τη διαδικασία ή για το ποιο θα είναι ο ρόλος ε, των αγροτών. Αν δεν έχετε αντίρρηση, αυτό θα κάνουμε. Προφανώς όταν γίνεται ενδιαφέρον το πράγμα και ζεσταίνεται η κατάσταση, μας πιέζει ο χρόνος, χρειάζεται χρόνος για να μας εξηγήσετε, ε, διαφωτίστε μας τα συγκεκριμένα ε, όσον αφορά τη σχέση με τη γεωργία, αλλά μην ε, μακρηγορήστε γιατί ακόμα έχουμε έξι ε, άτομα που ζητούν το λόγο και έχουμε και τις κυρίες Χάρκη. Ε, ε, κοιτάξτε, ορισμένοι από εμάς ε, ίσως να έχουν ερωτήσεις. Καλύτερα λοιπόν να κάνουμε πρώτα τις ερωτήσεις και μετά να ακούσουμε την απάντηση. Ε, κοιτάξτε, θα, έχετε, θα έχει χρόνο να απαντήσει. Πριν όμως ξεκινήσει η συζήτηση, νομίζω ότι είναι καλύτερα να ακούσουμε και τις δύο εισηγήσεις από τις δύο αρμόδιες γενικές διευθύνσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η παρουσία ήταν κοινή. Έτσι λοιπόν ο συνάδελφός μας από τη Γενική Διεύθυνση της Απασχόλησης κάλυψε και το θέμα της γεωργίας. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στη Γενική Αρχή. Γιατί να πρέπει να συμπεριληφθεί και η γεωργία σε αυτό το πακέτο. Ο λόγος ε, είναι παρεμφερής δηλαδή για να προσφέρουμε υποστήριξη σε όσους υποφέρουν από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης. Υπάρχει όμως και κάποια διαφοροποίηση, διότι μιλάμε για δύο διαφορετικούς τομείς. Καταρχήν, αναφερόμαστε στο γεγονός ότι δεν μιλάμε για αμοιβόμενους εργαζόμενους, αλλά για αυτοαπασχολούμενους που είναι οι περισσότεροι γεωργοί. Και δεύτερον, η δεύτερη μεγάλη διαφορά είναι ε, τα αίτια, πώς προκαλούνται όλες οι αρνητικές επιπτώσεις. Δηλαδή δεν έχουμε τόσο μεγάλες απολύσεις, διότι το τομέας είναι περισσότερο κατακαιρματισμένος. Κατά τα άλλα, ε, παρά τις διαφορές που υπάρχουν ε, και που πρέπει να ληφθούν υπόψη στον κανονισμό, στο πώς θα εφαρμοστεί ο στόχος είναι να είμαστε στοχευμένοι. Δηλαδή δεν μιλάμε εδώ για μία καταποκοπή αποζημίωση στη γεωργία. Ε, εκείνο που επιθυμούμε είναι να υπάρχει στοχευμένη υποστήριξη όπου οι γεωργοί οι οποίοι απασχολούνται σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ε, κάποιοι εξ αυτών επηρεάζονται περισσότερο. Αυτά σε γενικέ γραμμέ ήθελα να πω, αλλά όσον αφορά την πρώτη ερώτηση που ετέθη, μπορώ να σα εξηγήσω ακριβώ τι σημαίνουν αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν. Δηλαδή τα 4,8 δι ε, τη ζημιά, την απώλεια. Ε, αυτό είναι μια εκτίμηση αξιολόγηση. Υπάρχουν πολλά στοιχεία Ορισμένα εξ αυτών μόλις δημοσιεύτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει μια σειρά επιπτώσεων. Τα 4,8 εκατομμύρια, οι απώλειες ε, του, της Γεωργίας συγκρίνονται με την κατάσταση που υπήρχε χωρίς τη συμφωνία. Μιλάμε δηλαδή για το σύνολο των επιπτώσεων στο τέλος της προβλεπόμενης χρονικής περίοδου. Αυτά απλό για να σας διευκρινίσω τι ακριβώς σημαίνουν τα στοιχεία. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πώς, σε τι διαφέρει η διαδικασία. Όλοι ε, γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το EGF, τα κράτη-μέλη κλπ. Αλλά στην περίπτωση της Γεωργίας πώς λειτουργεί. Ωραία. Τότε θα μου επιτρέψει να αναφερθώ εν συντομία επ' αυτού. Ο συνάδελφός μου ανέφερε ότι ε, διαφέρει γιατί πρόκειται για μία ε, αντίδραση εκ των προτέρων και όχι εκ των υστέρων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των μισθωτών εργαζομένων. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Διότι δεν επιθυμούμε να περιμένουμε ο Γεωργός ε, να χάσει αν θέλετε τη δουλειά του πριν προβλέψει ο ίδιος να κάνει κάποια αλλαγή. Πώς μπορούμε λοιπόν να προτρέξουμε. Και το μόνο που γνωρίζουμε είναι σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση έχουμε μια επιχείρηση η οποία παραδείγματο χάρη αναθέτει σε εργολάβο στην Κίνα ή σε τρίτους ε, στην Κίνα ε, να παράγει να συνεργαστούν. Στη Γεωργία όμως γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι ε, ενεργοποιείται αυτός ο μηχανισμός της ε, παγκοσμιοποίησης. Γνωρίζουμε με βάση τις μελέτες μας ότι γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι ε, τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο. Μπορούμε λοιπόν να υποφεληθούμε από αυτές τις ε, πληροφορίες που έχουμε εκ των προτέρων για να προβλέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα μπορούμε. Και κάνουμε το εξής. μετά την θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας της εμπορικής συμφωνίας η Κομισιόν έχει κάποιο χρόνο πριν συζητηθεί η συμφωνία στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Εκείνη λοιπόν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Κομισιόν προβαίνει σε αξιολόγηση των επιπτώσεων και εντοπίζει τους ε, τομείς και τις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο. Με βάση αυτά τα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μια απόφαση όπου αναφέρει ποιοι θα είναι αυτοί οι τομείς, για ποιους τομείς μιλάμε και δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζουν τις αιτήσει τους. Όμως οι αιτήσει από τα κράτη-μέλη μπορούν να αποσταλούν μόνο εφόσον η συμφωνία έχει τεθεί σε ισχύ και μόνο εφόσον έχει προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στους γεωργούς. Αυτό είναι διαφορετικό από ε, την κανονική συμφωνία που ισχύει για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Όλα τα άλλα είναι τα ίδια ή μοιάζουν. Νομίζω ότι έτσι καταλαβαίνετε λιγάκι τη διαφορά ε, σε σχέση με την ενεργοποίηση. Πρέπει να λειτουργήσουμε ταχύτατα, να μην περιμένουμε ε, τις πρώτες επιπτώσεις για να δρομολογηθεί η όλη διαδικασία. Και νομίζω ή ελπίζω ότι σας έδωσα αρκετές εξηγήσεις από αυτού. Η κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, παρουσίασή της και θα ήθελα να ξεκινήσω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι ακόμα και μετά την εξήγηση που άκουσα το να συμπεριλαμβάνονται οι γεωργοί ε, σε διαφορετική βάση η γεωργία από ό,τι άλλοι τομείς αυτό κατά άποψή μου είναι γελίο θα το χαρακτήριζα. Υπάρχει εδώ ένα χάσμα σε σχέση με τον προεπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα των γεωργών. Εάν λοιπόν συμπεριληφθεί και η ιδέα του να αποζημιώνονται τομείς για νέες πολιτικές, δεν υπάρχει τέλος. Μπορεί κανείς ε, να αποζημιώσει ε, όλους τους τομείς ε, λόγω του ότι καλούνται να προβούν σε μέτρα αναδιάρθρωσης που να είναι φιλικά προς το περιβάλλον ή και πολλά άλλα μέτρα τα οποία έχουμε αποφασίσει. Άρα δηλαδή εδώ υπάρχει πραγματικός κίνδυνος. Και είτε θα πει κανείς ότι η γεωργία είναι ένας τομέας όπως όλοι οι άλλοι, δηλαδή αν κάποιοι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο μπορούν να είναι αποδέκτες αποζημίωσης, τότε ας πούμε μπορεί κανείς να πει εντάξει ας συμπεριληφθούν αυτοί. Αλλά το να προβλέπονται διαφορετικοί κανονισμοί για ένα τομέα, κατ' ουσίαν τι λέει κανείς. Λέει ότι θέλουμε ένα εργαλείο για να βοηθήσουμε τους ε, γεωργούς που έχουν προβλήματα και πού μπορούμε να βρούμε αυτά τα χρήματα. Α, ναι, πράγματι θα τα βρούμε από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Με λίγα λόγια, είτε για όλους ε, ε, τα ίδια, είτε καθόλου όχι να υπάρχει ξεχωριστή αντιμετώπιση της ε, γεωργίας. Επίσης, να σας πω κάτι, ότι μόλις γύρισα από ε, γονική άδεια, άδεια και πραγματικά ήταν το τελευταίο πράγμα αυτό που περίμενα να βρω μπροστά μου. Ε, σε τελική ανάλυση νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να βελτιωθούν σε σχέση με το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση που δεν έχουν αναφερθεί. Παραδείγματο χάρη, περίοδο εφαρμογή. Αναφέρθηκε η περίοδο αναφορά, αλλά όχι αυτή τη εφαρμογή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για πολλέ ε, περιπτώσει. Υπήρξε τουλάχιστον κατά το παρελθόν. Ή το πρόβλημα ότι πλούσιε χώρε, οι πιο πλούσιε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιμοποιούν περισσότερο το Ταμείο αυτό από ότι οι πιο φτωχέ. Κυρίω οι χώρε εκείνε οι οποίε αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα, αυτέ δεν δεν καταφεύγουν σε μεγάλο βαθμό στο ταμείο. Υπάρχουν λοιπόν στην Ελλάδα, παραδείγματο χάρη, πάρα πολλέ υπερβολικέ απολύσει, τεράστιε αριθμού απολύσεων και αυτοί δεν καταφεύγουν σε αυτό. Και εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι η συγχρηματοδότηση το πρόβλημα ή μήπω ε, το ότι δεν υπάρχει η διοικητική επάρκεια για να μπορέσει κανεί να ζητήσει αυτά τα κονδύλια. Το έχουμε ρωτήσει πολλέ φορέ και δεν μα απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μα είπε το πώ είναι δυνατόν το ότι οι φτωχότερε χώρε δεν κάνουν καλή χρήση αυτού του ταμείου, του εργαλείου. Και ένα από τα μεγαλύτερα ε, προβλήματα που έχουμε με το πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το Ταμείο είναι ότι οι πλούσιες επιχειρήσεις οι οποίες κάλλιστα μπορούν μόνες τους να αποζημιώσουν τους ε, απολυόμενους εργαζόμενους και αυτές μέσα από τους κανόνες είναι επιλέξιμες. Ε, εγώ θα έλεγα ότι η κρίση είναι μια πολύ πιο λογική βάση να εντάξουμε όλα αυτά από την παγκοσμιοποίηση. Γιατί αν μια εταιρεία, παραδείγματος χάρη, μετεγκαθίσταται σε μία τρίτη χώρα με χαμηλό κόστος μισθών. Πολύ συχνά οι εταιρείε αυτές έχουν αρκετή τη ε, ε, οικονομική επάρκεια για να μεριμνήσουν μόνες τους για τους απολυόμενους εργαζομένους. Εγώ πιστεύω ότι το Ταμείο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται περισσότερο κάτω από το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2020. Πώς μπορούμε δηλαδή να προσαρμοστούμε σε μια πιο πράσινη οικονομία, πώς μπορούμε να πάρουμε απολυόμενους εργαζομένους από απαρχαιωμένους ε, τομείς που δεν έχουν κανένα μέλλον και ίσως λόγω της παγκοσμιοποίησης, πώς μπορούμε αυτούς να τους μετεκπαιδεύσουμε, να ενταχθούν μέσα στη νέα οικονομία και πώς μπορούμε να βγούμε πιο ισχυροί και πιο πράσινοι από αυτή την κρίση. Αν έχει την καλοσύνη παρακαλώ θα ήθελα απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριος Νταρντέν και μετά κυρία Χάινερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχήν για την παρουσίαση που ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάποιες πρώτες σκέψεις μετά από αυτά που ακούσαμε. Χαίρομαι που υπάρχει ξεκάθαρη θέληση της Κομισιόν να ε, συνεχίσει, να διατηρήσει το Ταμείο αυτό, γιατί αδιαφυσβήτητα είναι χρήσιμο και απαραίτητο και αυτό το αποδεικνύει ο αριθμός των αυξανόμενων, ο αυξανόμενος των ε, ετοιμάτων. Παρενθετικά, αλλά και σημαντικά, υπάρχει η τρέχουσα συζήτηση για το σκέλος κρίση. Εκπλήσεται κανείς ότι δεν ε, έγινε δεκτή η πρόταση κάποιων κρατών μελών που θέλησαν να καταργηθεί ε, η δυνατότητα αιτήματος σε σχέση με την κρίση γιατί το, αυτό είναι το βασικό κίνητρο των αιτήσεων. Παρότι μπορεί κανείς να διαρωτηθεί πού βρίσκεται το ξεκίνημα της κρίσης σε σχέση με το ξεκίνημα της παγκοσμιοποίησης. Έχουμε την κρίση της κρίσης και την παγκοσμιοποίηση. Εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν μια παρένθεση θα επανέλθω σε λίγο. Θέλω, χαίρομαι λοιπόν που υπάρχει επιθυμία διατήρησης, είναι χρήσιμο ταμείο πρωτότυπο που βοηθά τους εργαζόμενους, ένα ταμείο που μπορεί να προσφέρει στην καταπολέμηση της φτώχειας, ένα θέμα που μας απασχόλησε την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλεια. Χαίρομαι επίσης για την παράταση που προτείνεται για το πεδίο εφαρμογή και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, σημαντικό. Και γιατί όχι και τους αγρότες. Νομίζω ότι ε, είναι ευχάριστη αυτή η ε, διεύρυνση παρότι έχει τα ανησυχητικά της. Όσον αφορά το κατόφλιο, επίσης είναι ενδιαφέρον ότι διατηρείται το, αυτό των 500 και όχι των χιλίων. θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα πιο κάτω και να συμπεριληφθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατ' εξαίρεση γιατί και όχι με πιο ανοιχτό τρόπο. Χαίρομαι επίσης για την ευελιξία όσον αφορά την τροποποίηση των τρεχουσών δράσεων. Ε, χρειάζεται λόγω της βραδίας επεξεργασίας. Χαίρομαι και για την αυξημένη τεχνική βοήθεια που προσφέρεται στα κράτη, γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολο να μπορεί κανείς να κινήσει τους κρατικούς μηχανισμούς. Με, ανησυχεί όμως, με ανησυχούν κάποια πράγματα. το μέρος που δεν έχει ε, ε απευθυνθεί στους, ε, ε, στους αγρότες. 500 εκατομμύρια για τα 5 χρόνια. Αυτό το θεωρώ αρνητική ένδειξη απέναντι ας πούμε στους εργαζόμενους στη βιομηχανία. Επίσης υπάρχουν υπάρχουν και κάποια θέματα που αφορούν τα κράτη για την ε, κρίση. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Και θα κλείσω κυρία Πρόεδρε λέγοντας ότι ε, δεν ξέρω τι να κάνω όσον αφορά τα μέτρα επιτάχυνσης της κινητοποίησης. Δεν υπάρχει στον κανονισμό. Και όσον αφορά την καθεστική ατάξη όσον αφορά το δημοσιονομικό καθεστώς του Ταμείου η εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων στην αρχή της υπόθεσης. Αυτό καμιά φορά δημιουργεί προβλήματα και παρατείνει τις προθεσμίες. Αν επιμείναμε σε αυτό, ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε το, να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα. Βλέπω ότι για τους αγρότες ε, κινούμαστε σε μια λογική του να προτρέξουμε. Το ίδιο ίσως θα έπρεπε να κάνουμε και για τους βιομηχανικούς εργαζόμενους. Αυτά, Πρόεδρος. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης έχει ε, πολύ καλή φήμη στην Αυστρία. Γιατί επιτέλους είναι ορατή η Ευρωπαϊκή Ένωση, εμφανίζεται ως πυροσβεστική θα έλεγα, πυροσβεστική υπηρεσία για να βοηθήσει τα θύματα της παγκοσμιοποίησης. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Ε, και έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά στους υποβάλλοντες αίτηση. Εσείς είπατε ότι μπορεί να είναι και δύο περιφέρειες. Εμένα με ενδιαφέρει να γνωρίζω κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει διασυνοριακά και αν ναι, ε, πρακτικά πώς εφαρμόζεται. Και κάτι άλλο σε σχέση ε, με αυτούς που χάνουν από τη Γεωργία λόγω των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών. Πρέπει να σας πω ότι πραγματικά είναι απίστευτο ε, σχεδόν δεν πιστεύω αυτά που ακούω, τις προτάσεις που υποβάλλονται. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρξει ε, μία άδικη μετατόπιση, η λαιλασία αν θέλετε, η φαρπαγή από για να δοθεί κάτι σε άλλους. Κοιτάξτε, η Γεωργία εδώ και χρόνια είναι θαυμάσια οργανωμένη και γι' αυτό λοιπόν είναι αδιανόητο γιατί ε, τα μέσα του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση δεν πρέπει να διατεθούν στη γεωργία. Α μην ξεχνάμε ότι εδώ ε, ποτίθεται ότι πρόκειται για ένα εργαλείο επίδειξη αλληλεγγύη, που σημαίνει δηλαδή ότι ε, θα υπάρχουν κερδισμένοι, αλλά θα υπάρχουν και χαμένοι. Και αυτά τα κονδύλια του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση υποτίθεται ότι προβλέπονται για τους χαμένους. Δεν θα πρέπει λοιπόν, όπως σας είπα, να υφαρπάξουμε από κάποιους ένα ποσό για να το μεταφέρουμε, να το δώσουμε σε κάποιους άλλους. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εμείς έχουμε υποβάλει σειρά προτάσεων για να βελτιώσουμε το Ταμείο με πρακτικούς τρόπους και περισσότερη δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν το πετύχαμε μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Όταν σοβεί κρίση σαν την παρούσα, όταν τα ποσοστά ενεργείας ε, έχουν φτάσει στα γνωστά επίπεδα, όταν οι εθνικοί προπολογισμοί δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της ανεργίας και για τη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών και της πρόνοιας, τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε αδυναμία να υποφεληθούν από ένα ταμείο σαν αυτό. Λόγω των διαδικασιών και των ορίων. Έχουμε παρακολουθήσει πολύ στενά την συζήτηση Ξέρουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις ε, έχουμε χώρες που πλήττονται από πολύ ψηλή ανεργία και δυστυχώς δεν μπορούν να υποφεληθούν από το Ταμείο. Λόγω πολλές φορές διοικητικών δυσκολιών, λόγω των διαδικασιών ή λόγω του ότι δεν έχουν τα ίδια τα κρατημέλη τα κονδύλια για να συγχρηματοδοτήσουν τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς είναι δυνατόν η Κομισιόν να ζητά συγχρηματοδότηση και μάλιστα υψηλότερη, λέει η μιλήτρια. Δεν καταλαβαίνω πού πηγαίνουμε. Τη στιγμή που η βασική φιλοσοφία του Ταμείου είναι να κινηθούμε με βάση κάποιες αρχές οι οποίες όμως βλέπω σήμερα δεν εξασφαλίζουν δικαιοσύνη και ισότιμη μεταχείριση. Τι θα κάνουμε με τους ανέργους στην Πορτογαλία. Για τους ίδιους ε, ανέργους, εμείς παίρνουμε 100.000 ευρώ, η Γερμανία σπράττει ένα εκατομμύριο. Αυτό αποτελεί αδικία. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί και γι' αυτό μια λύση. Η Κομισιόν έχει υποχρέωση να θεσπίσει διαφορετικούς κανόνες, διαφορετικούς κανόνες λειτουργίας του Ταμείου, έτσι ώστε το Ταμείο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι στις χώρες μας κατά τη διάρκεια αυτής της οξίας κρίσης. Δεν είναι δυνατόν τα κονδύλια του Ταμείου να πάνε στις πλούσιες χώρες τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τεράστιες δυσκολίες χωρίς να μπορούμε καν πολλές φορές να υποβάλουμε τις σχετικές αιτήσει. Αυτά είναι τα σχόλιά μου, αυτές είναι οι επικρίσεις μου και καλό συναφώς στην Κομισιόν να λάβει υπόψη τα προβλήματα αυτά για να προβεί στις αναγκαίες τροποποίησεις. Κάτι άλλο το οποίο μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι το θέμα της γεωργίας, της ένταξης των γεωργών. Κατά την άποψή μου, η κοινή αγροτική πολιτική έχει τα δικά της κονδύλια, τα δικά της εργαλεία, ας βρουν οι αγρότες εκεί τη λύση. Το λέω αυτό Χωρίς να διαφωνώ ότι χρειάζονται και οι αγρότες στήριξη. Δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό. Διαφωνώ όμως με τη χρήση του EGF για την υποστήριξη των αγροτών. Έχουμε αλλού ένα σωρό προβλήματα. Έχει φυσικά και η Γεωργία τα δικά της. Αυτά, κυρία Πρόεδρε. Αυτά είναι τα ζητήματα που ήθελα να θέσω και τα οποία θέλω να σκεφτεί η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, και έτσι κλείνει και ο κατάλογος των ομιλητών. Παρακαλώ. Κύριος Μπέκερ, ε, θα ήθελα να πω, για μένα είναι θετικό το γεγονός ότι τα κονδύλια του Ταμείου ε, προβλέπονται για ε, παροχή υποστήριξη σε περίοδο κρίσης και επίσης για να μην εκτραχυνθεί η κρίση. Ανταυτού από την άλλη πλευρά υπάρχουν βέβαια ξεκάθαρες δομές σε όλα τα ταμεία ε, και δεν ακούσαμε το τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά. Δεν ακούσαμε ολοκληρωμένο το σκηνικό και δεν ακούσαμε το πώς μπορεί να περιοριστεί η βοήθεια εις βάρος των υπολείπων. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα όπου κατά την άποψή μου δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσει κανείς αυτό το σκεπτικό. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχήν, όσον αφορά την παρουσίαση της πρότασης. Γιατί αν δούμε εδώ τα ποσά, θα έλθω στο θέμα σε λίγο. Το να υποστηρίσει κάποιος ότι το EGF επεκτείνεται και συμμελαμβάνει την γεωργία αποτελεί αντίφαση με την έννοια ότι δεν επεκτείνεται το EGF ε, στην Γεωργία. Η Γεωργία ε, θα έλεγα καταλαμβάνει το ίδιο το EGF. Δείτε τα νούμερα. Αν έτσι όντω έχουν τα πράγματα, νομίζω ότι δεν θα είμαστε πλέον εμεί ω Επιτροπή Αρμόδια για θέματα κοινωνική πολιτική. Είμαστε ανεφαντικημένου. Όσον αφορά τώρα το δικαστήριο και τις αποφάσεις του, πιστεύω ότι δεν πρέπει να χάσουμε μπροστά μας το πραγματικό διακύβευμα που είναι η κοινωνική πολιτική. Μετά είναι γεγονός ότι δεν έχουμε χρησιμοποιήσει επαρκώς τα κονδύλια του ταμείου, γιατί κάποιες χώρες δεν τα χρειάστηκαν, κάποιες άλλες δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες, δεν κατάλαβαν πώς λειτουργεί το ταμείο. Και είναι σαν να μας λέει κάποιος ότι τελικώς δεν χρειαζόμαστε το EGF και πετάμε τα λεφτά μας στην γεωργία. Τα τρία τέταρτα μάλιστα των κονδυλίων του ταμείου. Τελικά η παγκοσμιοποίηση θίγει ή όχι τη βιομηχανία μας. Μήπως δεν κατάλαβα καλά. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτά που μας προτείνετε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με βάση τα νούμερα που μας δίνετε τουλάχιστον. Μας είπατε για τη Συμφωνία Μερκοσούρ μας είπε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα επανέλθω στο θέμα σε λίγο. Όμως, όσον αφορά την κατανομή γεωργία, βιομηχανία, πραγματικά γιατί προβλέπουμε ήδη των προτέρων την κατανομή μεταξύ αυτών των δύο τομέων. Θα χρηματοδοτήσουμε όντως κοινωνικά μέτρα μέσω του EGF στην γεωργία Να πούμε τα πράγματα με το όνομά του σας παρακαλώ. Πρέπει να ικανοποιήσουμε από τη μια μεριά τα κρατημέλη, τα οποία δεν θέλουν να μειωθεί ο προπολογισμό τη Γεωργία και φοβούμαι ότι εδώ κάνουμε τι. Προσφέρουμε μέτρα υπό το κάλυμα, υπό το ένδυμα τη ε, κοινωνική πολιτική για να χρηματοδοτήσουμε την Γεωργία. Αυτό φοβάμαι ότι γίνεται. Αυτό παρακαλώ να το λάβει υπόψη η Κομισιόν. Πέρα μα λέτε ότι πρόκειται για κονδύλια για την αντιμετώπιση τη κρίση και γι' αυτό είναι εκτό προπολογισμού. Και τι να ισχύσει αυτό για τη Γεωργία. Μα λέτε την άλλη ε, στιγμή ότι ο κανονισμός προβλέπει ένα μόνιμο ταμείο. Έχουμε μια μόνιμη κρίση μήπως. Είναι μόνιμο το εργαλείο ή όχι λειτουργούμε σε μια ελεύθερη εσωτερική αγορά. Εδώ δεν πρόκειται για μετωπίση τη κρίση, φοβούμαι. Πρόκειται για μια νέα πολιτική. Μια νέα επιπλέον πολιτική. Δεν βλέπω, λοιπόν γιατί το Ταμείο παραμένει εκτός προπολογισμού. Όσον αφορά τώρα το ποσοστό συγχρηματοδότησης και παρέρχομαι και στα δικά σα άλλωστε συμπεράσματα και την ενδιάμεση αξιολόγηση. Ερωτώ, με βάση τα δεδομένα ποσοστά γιατί μια χώρα που έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Ταμείο συνοχή, γιατί να πάει στο EGF και όχι στο Ταμείο συνοχή. Δεν έχει κανένα απολύτω κίνητρο. Και το λέω αυτό γιατί αποσταθεροποιείται ακριβώς τα κράτη-μέλη τα οποία θα είχαν την δυνατότητα να προσφύγουν στο EGF, στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε το ποσοστό συγχρηματοδότησης να ποικίλει, να διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα και τις ανάγκες. Όπως ε, γίνεται με το Περιφερειακό Ταμείο, για παράδειγμα. Τώρα, όσον αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων ε, από τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Εδώ πραγματικά αρχίζω να μην καταλαβαίνω. Καταρχήν θέλω να μας δώσετε τα νούμερα, να δούμε την έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων. Ε, μας είπατε μείον 4,8 για τη Γεωργία, 8 συν 8 για τη βιομηχανία, συν 17 για τις υπηρεσίες. Ωραία, από αυτά τα δισεκατομμύρια που θα πάρει η Γεωργία, πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Σκεφτήκατε το άρθρο 9 της συνθήκης. Και τι γίνεται μετά συν 8 και συν 17 δισεκατομμύρια που πήγαν, αν, μιλάμε, αν θέλουμε να μιλάμε για κοινωνική πολιτική. Και ποια είναι τα δημοσιονομικά μέτρα, τα φορολογικά έσοδα ενδεχομένω που πετυχαίνουμε με το συν 8 και συν 17 δισεκατομμύρια. Η ερώτηση μου λοιπόν αφορά τις νέες θέσεις εργασίες που δημιουργούνται στην Ευρώπη και τα φορολογικά έσοδα. Τα ωφέλη για τον προπολογισμό. Και το θέμα της επανένταξης, τέλος, καταλαβαίνω το στόχο, αυτό που είπατε το 50% των εργαζομένων να επανενταχθεί. Πολύ καλό, καλό είναι να υπάρχει ένα όριο, μια λέξη απέτηση. Στην περίπτωση αυτή όμως, φοβούμαι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την ηλικία των εργαζομένων. Δείτε τι έγινε στην περίπτωση της Ρενό, τι έγινε στην Πορτογαλία, όταν ένα μέτρο εφαρμόζεται με τρόπο ισοπεδωτικό, με τον ίδιο τρόπο παντού. Θα μου πείτε, μας ενδιαφέρουν κυρίως οι εργαζομένοι που είναι τώρα στα 55 τους, για παράδειγμα. Όμως, η υλοποίηση ενός εξατομικευμένου προγράμματος για εργαζομένους που είναι 59, 60 ενδεχομένω. δεν νομίζω ότι θα μας επιτρέψει να πετύχουμε τους στόχους που θέτεται. Και το είδαμε και στην περίπτωση της Ρενό. Η υποθεμένη κατάρτιση όθησε ε, ανθρώπους να γίνουν ε, κυπουροί, ή να ασχοληθούν με ατομική περιποίηση και άλλους παράξενους τομεί. Σύμφωνα, βοηθούν αυτά τους ε, ανθρώπους να αντιμετωπίσουν ε, τη γύρανση και την έξοδο την αγορά Αλλά εδώ μιλάμε για ένα εργαλείο το οποίο με τις νέες δεξιότητες θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Δεν θα βοηθήσει την έξοδο στη σύνταξη. Μετά τα θέματα της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Ξέρω ότι εδώ δεν μιλάμε μόνο για την δημιουργία θέσεων εργασίες φυσικά, αλλά μια που αναθεωρούμε τον κανονισμό του EGF πρέπει να θέσουμε όλα τα θέματα στο τραπέζι. Συγγνώμη, ξέχασα και ένα σημείο πριν να μιλήσω για τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τι γίνεται με τους ε, πληθυσμούς στις περιοχές όπου γίνονται πωλήσει. Είπατε ότι συμπεριλαμβανομέν... συμπεριλαμβαν... θα συμπεριλάβουμε και τους ανεξάρτητους επαγγελματίε και τους επισυμβάσει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνεί. Ξέρω ότι πολλές μικρομεσαίες θίγονται από την παγκοσμιοποίηση και στον τομέα των, της υπεργολαβίας, στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, την υφαντουργία και ούτω καθεξής. Τώρα όσον αφορά, επανέρχομαι στον ρόλο του Κοινοβουλίου. Είτε πρόκειται για την βιομηχανία, είτε για την γεωργία, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφέρει τα μέγιστα. Είπε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας ότι μπορούμε να προβλέψουμε τις επερχόμενες καταστροφές στον τομέα της επασχόλησης στην ε, γεωργία λόγω των συμφωνιών που υπογράφουμε. Με συγχωρείτε, δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα σοφός κανείς για να καταλάβει ή να προβλέψει τι θα γίνει στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαντουργίας κλπ. Δεν ξέρω γιατί λοιπόν γιατί τόσο διαφορετικές είναι αυτέ οι δύο διαδικασίες, γιατί διαφοροποιείται τόσο πολύ ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αρτήση του αν πρόκειται για την γεωργία ή την βιομηχανία. Προκαλείται έτσι μια σύγχυση, κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι ο στόχος που επιδιώκουμε. Έχω σχόλια λοιπόν και για το Συμβουλίο και την Κομισιόν. Αναγνωρίζω βεβαίω την πρώτη φορά που συζητούμε το θέμα αυτό εδώ στην Επιτροπή μας, ε, εξαιρετικά σημαντικό το θέμα. Να δώσω όμω τον λόγο στον κύριο Λεμπρά. Ε, δεν ξέρω, έχουμε πέντε λεπτά από τους Δερμηνείς για να ε, ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους βουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ και να απαντήσω όσον αφορά την εξαίρεση λόγω κρίση. Η Κομισιόν μαζί με το Κοινοβούλιο ανησυχεί για την στάση του Συμβουλίου. Και θα ξαναπώ ότι θα ήταν παράλογο να δεχτούμε ότι η κρίση τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2011. Ανησυχούμε, όπως καταλαβαίνετε, και εμείς όπως και εσείς. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση δύο ή περισσότερων περιφερειών σε ένα πρόγραμμα ε, και το θέμα της ε, συγχρηματοδότησης. Όπως προείπα, εάν η βασική συγχρηματοδότηση είναι 50%, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ανέλθει σε 65% για περιοχές στις οποίες υπάρχουν ακόμη πιο μεγάλες δυσκολίες. Από εκεί πέρα, είμαστε έτοιμοι να επιδείξουμε ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία να διαφοροποιήσουμε θα έλεγα τα ποσοστά συναρτήση της χώρας στόχου, δηλαδή 50% για τις πλούσιες χώρες, 65% για τις πιο φτωχές. Θυμίζω για την ιστορία, όσον αφορά την εξαίρεση λόγω κρίσης το 2009, η Κομισιόν είχε προτείνει 75% ποσοστό χρηματοδότησης και αυτό το σταμάτησαν στο Συμβούλιο, το 75%. Αν δείτε τώρα που βρισκόμαστε σήμερα, με την παράταση της εξαίρεσης λόγω κρίσης, ε, το ότι πετύχαμε το 65%, φοβούμαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την νέα προγραμματική περίοδο να ξεπεράσουμε, να υπερβούμε το 65% λόγω Συμβουλίου. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της ισότιμης μεταχείρισης που θίξετε, είναι σαφές ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της προσφυγής στο EGF, στο ταμείο μας, από την μια μεριά, όσον αφορά την χρηματοδότηση αναεργαζόμενο, αν συγκρίνεται δηλαδή ε, την Πορτογαλία με την Γερμανία. 2.000 για την Πορτογαλία, 5.000 για την Γερμανία. Και αυτό είναι απλώς διονδεικτικά νούμερα. Αυτό ισχύει. Είναι όπως το είπατε. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε γιατροί χωρίς σύνορα. Δεν καθορίζουμε εμείς τα μέτρα. Τα μέτρα τα καθορίζουν, τα προτείνουν και τα καθορίζουν τα κράτη-μέλη με βάση την δική τους εμπειρία, τα εθνικά συστήματα, την κατάσταση στη χώρα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και θεσπίσαμε τον στόχο του 50% όσον αφορά την επανένταξη των εργαζομένων δηλαδή, για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν τα προγράμματα τα οποία θεωρούν ότι έχουν πιθανότητες επιτυχίας. Γι' αυτό και θέσαμε και το ανώτατο όριο του 50% όσον αφορά τα λεγόμενα παθητικά μέτρα για τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την ε, ισότιμη μεταχείριση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απολαύουν ίδιες μεταχείρισης με τις μεγάλες. Μπορούμε πλέον να παρέμβουμε και σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε τομεακό. Τρεις είναι οι τρόποι παρέμβασης του Ταμείου. Μπορούμε να παρέμβουμε στην περίπτωση μιας μεγάλης επιχείρησης και των υπεργολάβων της. Μπορούμε να παρέμβουμε σε εξαιρετικέ περιπτώσεις, σε μικρές αγορές ή σε έναν τομέα ή σε μια περιφέρεια. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να κάνουμε πολλά πράγματα και για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει που μπορεί να είναι και οι προλάβει σε μεγάλε επιχειρήσει. Λαμβάνουμε υπόψη μα και θέλουμε επιλέξουμε πλέον του ιδιοκτήτες ε, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη διάρκεια αυτή τη μεταβατική φάση. Αυτά με την ελπίδα ότι απήντησα σε αρκετές από τις ερωτήσεις σας. Να δω αν ξέχασα κάτι. Θα αφήσω τους ε, συναδέλφους να απαντήσουν όσον αφορά τα θέματα της γεωργίας. Πιστεύω πάντως ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να επιταχύνουμε τις σχετικές διαδικασίες στο μέτρο του δυνατού. Όμως δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι επί της ουσίας το Ταμείο παραμένει εκτός προϋπολογισμού και το εξήγησε προηγουμένως αυτό έγινε επειδή δεν θελήσαμε να κρατήσουμε στην άκρη έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Να πούμε για παράδειγμα 350 εκατομμύρια το χρόνο και να τα προσθέσουμε στον προϋπολογισμό. Γιατί μπορεί μια χρονιά να χρησιμοποιήσουμε μόνο 50 εκατομμύρια, τα 300 να μείνουν αχρησιμοποιητά. Γι' αυτό κρίναμε πιο χρήσιμο να συνεχίσουμε να κινούμεθα εκτός προπολογισμού για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα διαθέσιμα περιθώρια και να μεγιστοποιήσουμε την αξιοποίηση αυτών των κοινοτικών κονδυλίων. Η διαδικασία αυτή θα κρατήσει, είναι βέβαιο. Όμω τουλάχιστον επιταχύνουμε τι διαδικασίε. Τα κρατη έχουν περισσότερη πείρα τώρα. Γνωρίζουμε και εμεί καλύτερα τα εθνικά συστήματα και εμεί επιταχύνουμε τη δική μα εργασία. Μπορεί να υπάρχουν καλύτερες διαδικασίες, δεν λέω, αλλά στην επόμενη σύσκεψη του EGF θα καταθέσω προτάσεις, έστω και άτυπα, για τη βελτίωση των διαδικασιών. Μπορούμε να επιταχύνουμε περαιτέρω τις διαδικασίες, ε, γιατί είναι προφανές ότι χρειάζεται όπου επεμβαίνουμε να παρεμβαίνουμε ταχύτατα. Πρέπει όμως και τα κράτη-μέλη να κάνουν τη δική τους δουλειά, ώστε η συγχρηματοδότηση να ακολουθήσει. Πρέπει να σας πω ότι σε καμία περίπτωση δεν χάσαμε πόρους. Κανείς δεν έχασε πόρους από το EGF. Χάρη στη συνεργασία όλων και με εσά. Δεν χάθηκε, επαναλαμβάνω, καμία αίτηση. Όλες ικανοποιήθηκαν γιατί σε άλλε περιπτώσει, σε άλλα ταμεία, σε άλλε παρεμβάσει έχουμε και ποσοστά 70% αποτυχία. Λοιπόν, θέλουμε να παρεμβαίνουμε, όχι το αντίθετο. Όμω, η πρωτοβουλία, θυμίζω, στι περιπτώσει μαζικών απολύσεων είναι στα χέρια των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη υλοποιούν τα μέτρα. Εμεί θα είμαστε αλληλέγγυοι και θα συγχρηματοδοτήσουμε. Θα διευκολύνουμε φυσικά την ανταλλαγή καλών πρακτικών, αλλά το ξαναλέω, η κύρια ευθύνη, η πρωτοβουλία είναι στα χέρια των κρατών μελών. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή με την εξαίρεση λόγω κρίση, γιατί ξεκινήσαμε από την παγκοσμιοποίηση, που είναι ένα γενικό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα επιδείξουμε αλληλεγγύη. Όμω, όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε την ε, κρίση, κάποια κρατημέλη λένε «Α, η κρίση είναι υπόθεση συγκεκριμένων κρατών μελών και όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να πίνησα, κυρία Πρόεδρε. Ξέρω ότι ο χρόνο πιέζει. Ε, ο λόγος στον ε, συναδελφό μου από την Γενική Διευθύνση Γεωργίας για να απαντήσει στι άλλε ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, εξαιρετικά χρήσιμα. Θα ήθελα να αναφέρω ένα βασικό ζήτημα πλέον. Ε, να σας πω ε, γιατί θελήσαμε αυτό τον ε, κανονισμό. Ε, έχουμε λοιπόν αυτή την εντολή από τον προϋπολογισμό και ήταν αρκετά τολμηρό το να επεκτείνουμε την υποστήριξη και στους γεωργούς ε, θύματα της ε, παγκοσμιοποίησης. Συνδυάζοντας αυτά με την πρόταση για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, κατέστη δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο δυνατότητες από κοινού. Και προτείνουμε κάτι το οποίο δεν είναι περιοριστικό είναι ένα ταμείο το οποίο ενεργοποιείται όταν υπάρχει συμφωνία, όταν υπάρχει αύξηση των εισαγωγών, μείωση των τιμών. Δεν πρόκειται λοιπόν για καταποκοπή αποζημίωση για όλους. Είναι στοχευμένη και μετά είναι υποστήριξη για να βοηθούν, βοηθηθούν οι γεωργοί να προσαρμοστούν, να αλλάξουν. να βγουν από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία ε, εμπίπτουν. Τώρα, σημείο 5 που αφορά τη γεωργία. Δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο η γεωργία θα χρησιμοποιεί αυτό το 2,5 ακόμα και στην ε, περίπτωση που υπάρξει μια εμπορική συμφωνία για πάρα πολλά χρόνια ενδέχεται το Ταμείο να μην χρησιμοποιηθεί για τον γεωργικό τομέα. Και μετά όσον αφορά τις ε, μελέτες ε, επιπτώσεων, αξιολόγηση επιπτώσεων. Οι τελευταίε που δημοσιεύτηκαν την ε, προηγούμενη εβδομάδα είναι πολύ πιο λεπτομερεί στι ε, περιφερειακές επιπτώσει ε, και μπορούμε να γνωστοποιήσουμε στη γραμματεία το link που υπάρχει για να μπορεί κανεί να μπαίνει και να παίρνει τι απαραίτητε πληροφορίε. Εκεί περιλαμβάνονται πληροφορίε για τι επιπτώσει στη γεωργία, στην παροχή υπηρεσιών και στη βιομηχανία. Όταν λέμε βιομηχανία μιλάμε για ένα πολύ ευρύ τομέα. Υπάρχει και εκεί υποδιέρεση σε διάφορους υποτομής και γίνεται και ποσοτικοποίηση ε, το θέμα της απασχόλησης και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο εξωτερικό. Θα δείτε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, διαφορετικές μελέτες, δίστανται και οι απόψεις. Ε, εντάξει, στη γενική κατεύθυνση ε, συμπίπτουν οι απόψεις, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και διαφορές. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για σήμερα. Πρώτος ευχαριστή και τους Δερμήνες. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα τα ξαναπούμε στις 5 Δεκεμβρίου το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.